Ε, Καλημέρα σα. Συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Στην πραγματικότητα υπήρξαν διάφορα πρακτικά προβλήματα. Το αυτοκίνητο που ε, έπρεπε να έρθει να με πάρει καθυστέρηση καθυστέρηση, έπρεπε να βρω εναλλακτική διαδρομή και υπήρχε τελικά περισσότερη κίνηση και έγιναν τα πράγματα χειρότερα. Γι' αυτό συζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα και μάλιστα στη συνεδρίαση στην οποία προεδρεύω εγώ η ίδια. Ζητώ συγγνώμη και από τους Δερμηνείς και από τη Γραμματεία. Θα ήθελα να έχουμε κάποιες εξηγήσει από τους συναδέλφους που πήγαν στο Μπαγκλαντές, να μας πούν λίγα λόγια για την αποστολή τους. που σιάζουν, να δώσω το λόγο στον κύριο Γιώσεφ Βαντενχόλσερ για να ξεκινήσει, αν είναι έτοιμος, για να μας εξηγήσει για την αποστολή στο Μπαγκλαντές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βαντενχόλσερ. Να σας πω για την ε, αποστολή το Μπαγκλαντές. 16 με 20 Φεβρουαρίου την περασμένη εβδομάδα πήγαμε στην Τάκα. Ήταν πάρα πολύ τεταμένα τα πράγματα από πλευράς ασφαλείας και η κατάσταση δυστυχώς έχει πάρει την κατηφόρα. Πάνε πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Η προετοιμασία της αντιπροσωπείας ήταν πάρα πολύ καλή. Από τη δική μας αντιπροσωπεία εκεί, ο Πιέρ ο δικός μας ε, πρέσβης είχε προετοιμάσει τα πάντα και μας συνόδευε συνεχώς. Θέλω να ευχαριστήσω και τη γραμματεία. Ήταν πάρα πολύ άρτια η ε, προετοιμασία και πάρα πολύ καλή. 23 παρακαλώ συναντήσεις είχαμε με διαφόρους. Ήταν πάρα πολύ εντατικό ε, το ταξίδι αλλά δεν πήγαμε στα πιο επικίνδυνα μέρη λόγω της κατάστασης της ασφαλείας. Λοιπόν, ποιο ήταν το κέντρο βάρους μας. Ε, τι θέλαμε να κοιτάξουμε. Φυσικά τα τραγικά γεγονότα πριν από δύο χρόνια στη Ράνα Πλάζα. Θυμάστε ότι κατέρευσε ένα εργοστάσιο και πέθαναν χίλιοι άνθρωποι. Γι' αυτό πήγαμε να δούμε επί τόπου πώς έχει η κατάσταση ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως των εργασιακών ε, διαπιστώσαμε χωρίς καμιά αμφιβολία ότι με το πρόγραμμα Accord έχουν γίνει κάποιες σημαντικές βελτιώσεις. Η ασφάλεια στην εργασία έχει αυξηθεί, ε, έχουν κάποια στοιχειώδη συνεννόηση των τέρων. Ε, τα συνδικάτα βέβαια καταλαβαίνετε ότι είναι υποτυπώδη και δεν ε, ανταποκρίνονται σε αυτό που θα έπρεπε. Πάντως πρόοδοι έχουν γίνει και σημαντικές και και ορατές. Ασχοληθήκαμε και με τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ελευθερία της έκφρασης. Ε, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ αφηρό μηδιακό τοπίο, ε, πάρα <laughs> πολλούς σταθμούς και κανάλια, αλλά μας είπανε ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι υπάρχει ελευθεροτυπία. Παραμένει το θέμα της ελευθερίας των μέσων να προξενεί ανησυχία. Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα είναι η νομοθεσία για τις ε, ξένες ε, δωρές, foreign donations, για ΜΚΟ από το εξωτερικό, θα ελέγχονται πιο αυστηρά από χώρες όπως η Ρωσία και άλλες ε, ακούμε αντίστοιχα επιχειρήματα και επιμείναμε πάρα πολύ ότι δεν γίνεται αυτό. Είναι ε, σημαντική επιδείνωση και επιβάρυνση των δυνατοτήτων ε, εργασίας των μη κυβερνητικών οργανώσεων που είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στο Παγκλαντές και δεν πρέπει να εμποδίζεται η δουλειά τους. Μας είπαν ότι ναι, αλλά εμείς θέλουμε να πατάξουμε την ε, τρομοκρατία γιατί μπορεί να χρηματοδοτείται με αυτούς τους διάβλους. Τα ακούμε αυτά τα επιχειρήματα και από συζητήσεις με άλλες χώρες όπως σας είπα. Τους είπαμε για τη θανατική ποινή και εξακολουθούμε να τονίζουμε ότι είναι απαράδεκτο από ευρωπαϊκή σκοπιά. Και παρακολουθούμε την κατάσταση από πάρα πολύ κοντά. Και με το Διεθνές ε, Δικαστήριο θα πρέπει ε, να εφαρμοστούν οι σχετικές νομοθεσίες και τα όσα αφορούν τα γεγονότα του 1971. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ε, η αναγκαστική γάμη ε, σε πολύ νεαρή ηλικία, πολύ μικρά κορίτσια υποχρεώνονται παντρεύονται και ε, βέβαια έχουν γίνει μεγάλες πρόοδοι και μεγάλα βήματα πρόοδου ε, στα γυναικεία δικαιώματα αλλά δεν έχει λήξει. Σας τα λέω επί τώρα. Ε, επίσης υπάρχει και το θέμα των αυτοχθόνων ε, μειονοτήτων έχουν θέμα εκεί με το αν θα του χαρακτηρίζουν αυτόχθονες, indigenous ή όχι. Γιατί αυτό έχει να κάνει και με θέματα ιδιοκτησίας. Και ένα από τα συμπεράσματα για μας θα πρέπει να είναι το θέμα της υφαρπαγής ε, γης, land grabbing, όχι μόνο στο Μπαγκλαντές γενικότερα. Και ένα τελευταίο. Ή ο Χίνκας. Που ε, το υποτιμούν οι αρχές ε, της χώρας ότι καλά εντάξει δεν είναι και κανένα ε, σημαντικό θέμα. Να μπορεί να προκύψει όμως, γιατί αν αυξηθούν οι μεταναστευτικές ροές ε, ε, θα υπάρξει επιβάρυνση τα σύνορα. Σας είπα ότι υπάρχει θέμα ασφαλείας από τις 5 Ιανουαρίου όπου συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τις εκλογές γίνονται ταραχές πάνω από 60 είναι νεκροί. 7 με 10 χιλιάδες ακούσαμε ότι ε, οπαδοί της αντιπολίτευσης έχουν συλληφθεί και φυλακιστεί. Η ίδια κυβέρνηση θεωρεί ότι έχει εκλεγεί νόμιμα και ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές με την αντιπολίτευση και είναι δύσκολο να λυθούν αν εμένουν ε, και οι δύο στις θέσεις αυτές. και όλα αυτά βασίζονται σε κάποια αποθυμένα του παρελθόντος. Δεν υπάρχει ούτε καν σε λεκτικό επίπεδο κάποια προσπάθεια κατευνασμού. Είναι όλα πάρα πολύ ε, άκαμπτα και ανένδοτα. Και με τον Μοχάμετ Ιουνούς είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με ε, δημοσιογράφους και εκπροσώπους της εθνούς κοινότητας και όλοι έχουν την ίδια εκτίμηση. Αν δεν αλλάξει τίποτα τις επόμενες εβδομάδες μπορεί να οξυνθεί ε, ακόμα περισσότερο κατάσταση μέχρι και εμφύλιο πόλεμο να έχουν. Όπως και να εξελιχθούν τα πράγματα, η προσωπική μου άποψη είναι αν το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πατάξουν την ίν αντιπολίτευση PNB, αυτό θα σημαίνει ότι θα υπάρξουν άλλες δυνάμεις που περιμένουν ή και καραδοκούν να προσφύγουν ακόμα και σε τρομοκρατία. Και ο μεγάλος κίνδυνος τώρα στο Βαγκλαντές είναι αυτός. Είναι, ξέρετε, μουσουλμανική χώρα, σπουδαία, καταπληκτική, αλλά υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Μέσα σε λίγους μήνες δηλαδή να ε, ε, δημιουργηθεί, να καλλιεργηθεί το έδαφος για να επικρατήσουν εξτρεμιστικές ομάδες. Που δεν τις θέλουμε ούτε εμείς ούτε η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές. Γι' αυτό θα πρέπει να ασχοληθούμε πιο εντατικά με τη χώρα αυτή, να την προσέξουμε περισσότερο. Και χτες ε, λύπη μας διαπιστώσαμε ότι εκδόθηκε ε, ένταλμα σύλληψης που δεν έχει ακόμα εκτελεστεί κατά τη ηγέτηδας της αντιπολίτευσης. Και ξέρουμε και ε, ότι συνελήφθηκε κάποιος που συναντήσαμε ε, στη συνεδρίαση που είχαμε μαζί της. Αυτό δεν είναι τρομερή όξυνση. Εάν συλληφθεί η Σακαλέντα, βέβαια οι λόγοι είναι θέματα διαφθοράς και τέτοια. Αλλά ε, εάν φυλακιστεί θα ε, είναι κάτι αυτό που θα οξύνει πάρα πολύ τα πράγματα. Αυτά όσο γινόταν πιο γρήγορα, σας είπα για τους Ροχίνγκας, για την αντιπολίτευση κτλ. Ε, ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώσεφ. Ο κύριος Κάρσκι, που ήταν επίσης μέλος της ε, αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι μετά από την πολύ λεπτομερή έκθεση του Γιώζεφ, σίγουρα δεν υπάρχουν και πολλά να προσθέσει κανείς. Ωστόσο, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω θερμά τη γραμματεία και την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ντακάρ. Και η Γραμματεία και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν οργανώσει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Είχαμε 23 συναντήσεις με προσώπους κυβέρνησης, αντιπολίτευσης, ε, συνδικαλιστικών οργανώσεων, ε, οργανώσεων της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, ε, με δημοσιογράφους μεταξύ άλλων. Ήταν πολύ εντατικό λοιπόν το πρόγραμμα και αυτό ήταν καλό διότι μας επέτρεψε να αποκτήσουμε συνολική εικόνα για το τι συμβαίνει στον Παγκλατές αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να προσθέσω ακόμη ότι αυτό που μας ενδιέφερε κυρίως ήταν τα εργασιακά δικαιώματα, τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και στο Μπαγκλαντές ε, ξέρετε, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα συνδικαλιστικά σωματεία είναι πάρα πολύ ε, ασθενή, πάρα πολύ αδύναμα. Μόνο το 2% των ε, εργαζομένων είναι μέλος συνδικαλιστικών οργανώσεων. Δεν είναι ένα μοντέλο που μπορεί να ενισχύσει τα εργασιακά δικαιώματα και ούτε καν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το δικαίωμα στην ασφάλεια στο χώρο εργασίας, την απαγόρευση απασχόλησης παιδιών που θα εργάζονται, π.χ. στην κλωστοϊφαντουργία, μεταξύ άλλων. Παρ' όλα αυτά, κάποια πρόοδος έχει σημειωθεί και είναι ορατή. Τους τελευταίους μήνες είδαμε αύξηση στον αριθμό καταχώρησης ε, σε επίσημους καταλόγους νέων συνδικαλωστικών οργανώσεων που συστάθηκαν. Και ελπίζουμε να αυξηθεί ε, η παρουσία μελών στα συνδικάτα όλο και περισσότερο. Η τάση δηλαδή έχει θετικό πρόσημο. Κάτι άλλο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι τα θετικά προγράμματα που εφαρμόζονται και υλοποιούνται στο Μπαγκλαντές σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορέσαμε να ε, εστιάσουμε την προσοχή μας, να δούμε ένα, την υλοποίηση ενός προγράμματος από κοντά, ενός προγράμματος που έχει σημείο εστίαση στα παιδιά. Υπήρχε ένα πρόγραμμα δηλαδή για να έχουν τα παιδιά ταυτότητα, έγγραφα πιστοποίηση της ταυτότητάς τους. Γιατί αν δεν υπάρχουν έγγραφα πιστοποιητικά γέννηση ή ταυτότητας, ο άνθρωπος, το ανθρώπινο όν δεν υπάρχει επισήμως. Και Εάν διατρέξουν ε, κίνδυνο, είναι πιο εύκολο να αναγνωριστούν. Τα παιδιά έτσι δεν θα είναι ανώνυμοι. ανώνυμα. Μας είπαν τα μέλη της ε, οργάνωσης αυτής ότι όταν μιλούν στην αστυνομία και βλέπουν ότι τα παιδιά έχουν έγγραφα που να πιστοποιούν την ταυτότητά τους, τότε αισθάνονται καλύτερα και τη χάνουν καλύτερης μεταχείρισης. Και θα θέλαμε όλα αυτά να τα ε, μεταφέρουμε αυτά που γίνονται στον Ντακάρ να τα μεταφέρουμε και αλλού σε αυτή τη χώρα των 160 εκατομμυρίων ε, στην Τάκα με συγχωρείτε ε, στη χώρα αυτή των 160 εκατομμυρίων κατοίκων και τέλος να αναφερθώ στα δικαιώματα των γυναικών από τη μία πλευρά Η γυναικεία παρουσία γίνεται όλο και πιο ισχυρή ε, στα υψηλότερα αξιώματα της διοίκησης στη χώρα. Η Πρωθυπουργό τη χώρα είναι γυναίκα και ενώ είναι μουσουλμανική χώρα. Η αρχηγό τη αντιπολίτευση είναι γυναίκα και η πρόεδρο του Κοινοβουλίου είναι γυναίκα. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι δεν υπάρχουν επιφυλάξεις ως προς τα, ε, το να ε, δώσουν σε γυναίκες τα υψηλότερα αξιώματα ε, της χώρας αυτής. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι Οι διεθνείς συνθήκες ή συμβάσεις για τα δικαιώματα των γυναικών θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως και αυτό πρέπει να επισημαθεί ε, στις αρχές του Μπαγκλατές. Το Μπαγκλατές είναι συμβαλόμενο μέρος στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των γυναικών. Ωστόσο, είναι μία από τις χώρες που έχει εκφράσει επιφυλάξει για τη σύμβαση αυτή καθεαυτή. Ως εκ τούτου, όταν ε, ασχοληθούμε ξανά με το θέμα αυτό, θα πρέπει να δράξουμε κάθε ευκαιρία για να επισημάνουμε στις αρχές του Μπαγκλαντές την ανάγκη να αποσύρει αυτή την επιφύλαξη έτσι ώστε το πλήρες περιεχόμενο της ε, ε, σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των γυναικών να μπορέσει να εφαρμοστεί στην πράξη. Ε, η αποστολή λοιπόν κύλησε πολύ εντατικά. Είχαμε 23 συναντήσεις σε τρεις μέρες. Προσγειωθήκαμε στις 5 και μισή και η πρώτη μας συνάντηση ήταν ήδη προγραμματισμένη για τις 8, δυόμιση ώρες μετά. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Επομένως έχετε ε, πραγματικά ε, κάνει να ακουστεί πολύ δυνατά η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Μπαγκλαντές και αυτό είναι καλό για το δικό μας ε, Κοινοβούλιο. Ο κύριος Τάνο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο φορές στη μετάφραση ε, υπόθηκε ότι το Μπαγκλαντές είναι μουσουλμανική χώρα, αλλά δεν είναι. Είναι κοσμική χώρα με κοσμικό σύνταγμα όπου οι μουσουλμάνοι είναι πλειοψηφία στο πληθυσμό. Αυτό έχει διαφορά. Ξέρετε, πριν από έξι χρόνια είχα συμμετάσχει σε μία αποστολή παρατήρησης των εκλογών. Πρέπει να σας πω ότι έχει τεράστια διασπορά, ομογένεια, παρόντες πάρα πολλοί Μπαγκλεντεσιανοί, π.χ. στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο και άρα γι' αυτό εγώ έχω ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο να καταλάβω ακόμα καλύτερα αυτή τη χώρα. Θα ήθελα να ε, ρωτήσω κάτι τον επικεφαλής της αποστολής που παραπονέθηκε για το ε, σχέδιο για τις ξένες δωρεές θα πρέπει να, και συνεισφορές. Θα πρέπει να κάνουμε την αναλογία με τη Ρωσία. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει σύγκριση. Η Ρωσία αποκλεί της ε, ΜΚΟ για να μην υπάρξει δημοκρατία στη χώρα αυτή. Το Μπαγκλαντές όμως δυστυχώς εξαναγκάστηκε να περιορίσει τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ. Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο. Το Μαγκλαντές είναι πολύ ευαίσθητη χώρα, εύθραυστη, πάρα πολύ ο πληθυσμό, πάρα πολλά προβλήματα με την υγεία, με την ασφάλεια, με την εργασία, στα εργοστάσια, παιδική εργασία και ούτω καθεξής. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα προβλήματα και θέλει να τα λύσει. Και ε, δυσκολεύεται ιδιαιτέρως γιατί ένα πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση των ε, ε, άκρο ισλαμιστικών οργανώσεων οι οποίες χρηματοδοτούν το κόμμα Τζαλάμ είναι ε, ε, σαλαφιστές και είδα πολιτικούς του Τζαμάτ με πολύ καλή χρηματοδότηση και δικηγόρους αντίστοιχα να υπερασπίζονται τους εγκληματίες πολέμου που κατηγορούνται για τις φρικτές βιοπραγίες του αγώνα απελευθέρωσης της χώρας του 1971. Δηλαδή πρέπει να παρεμποδίσουμε τη ροή του χρήματος από τη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ. Πρέπει να προλάβουμε έτσι ώστε να μην υπάρξει τεράστια απόλωση και ρίζος ριζοσπαστικοποίηση μιας χώρας η οποία ε, ήταν κυρίως υπέρ του σουφισμού, η οποία ήταν αρκετά μετριοπαθής και δεν θα πρέπει να γίνονται συγκρίσεις μεταξύ ε, της κυβέρνησης του Μπαγκλαντές και ε, το, της κυβέρνησης Πούτιν στην Ρουσία. Η διαφορά είναι τεράστια. Ε, οι προκλήσεις του Μπαγκλαντές είναι πολύ διαφορετικές, πάρα πολύ σημαντικές. Θα πρέπει να στηρίξουμε τον Μπαγκλαντές. Είναι μια χώρα στρατηγικής σημασίας για εμάς. Είναι ένα μοντέλο για την εκπαίδευση των γυναικών, για την ισότητα των γυναικών και ανδρών Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά συνήθιστο στον Ισλαμικό κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ για τα σχόλιά σας και τις σκέψεις σας και επειδή συμπληρώσατε την οπτική επί του Μπαγκλατές, εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε και μια γραπτή ενημέρωση για την αποστολή για να μπορούσαμε να εργαστούμε από τους βουλευτές και από τη γραμματεία που ταξίδεψαν εκεί. Όμως, ε, εγώ θα ήθελα να έχουμε μια γραπτή έκθεση στα πρακτικά της Επιτροπής μας από κάθε μετακίνηση. Έτσι λοιπόν, ε, θα ζητούσα από τους υπεύθυνους του Γραμματεία που έκαναν εξαιρετική δουλειά στην προετοιμασία της αποστολής και από τους βουλευτές που συμμετείχαν, αν θα μπορούσαμε να έχουμε μια γραπτή έκθεση σχετικά με την αποστολή. Παρακαλώ, ο κύριος Κάσκη. Θέλετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Για να αποφύγουμε κάποιες παρεξηγήσεις, εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω με τον κύριο Τάνοκ, ε, φοβάμαι, αν ε, και προερχόμαστε την διαπολιτική ομάδα. Δεν ξέρω, μήπως ε, υπήρχε και κάποια παρανόηση. Είτε είναι μουσουλμανικό κράτος ή όχι, Φυσικά δεν συμφωνώ ότι είναι σημαντικό το Σύνταγμα και όσα λέγονται στο Σύνταγμα είναι σημαντικά. Παρ' όλα αυτά, όταν ε, εγώ συνομίλησα με τους εκπροσώπους ε, των εθνοτικών μειονοτήτων και των θρησκευτικών μειονοτήτων, υπάρχει κάποια επικάλυψη φυσικά και μπορώ να δω μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα στην πράξη. Πρόκειται για μια χώρα η οποία περιγράφεται ως μια χώρα όπου η κρατική θρησκεία είναι το Ισλάμ. Οι ορτασμοί, οποιοδήποτε επίσημος εορτασμός έχει αυτό το χαρακτήρα. Αυτό είναι το ένα. Επίσης, έγινε λόγο σύγκριση του ρωσικού μοντέλου με το κλαντεσιανό μοντέλο σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της ε, της χρηματοδότησης. Προφανώς ε, δεν είναι η ίδια η κατάσταση σε κάθε χώρα. Πράγματι, υπάρχει ένας γενικός κανονισμός στο Μπαγκλαντέ. σε σχέση με τις ροές χρηματοδότησης από το εξωτερικό τις καθίστα κάποιος πιο δύσκολες. Διάφοροι δωρητές μας είπαν ότι η χρηματοδότηση των ΜΚΟ θα είναι πολύ δύσκολη. Βρίσκονται σε μια κατάσταση νομικού κενού. Οποιαδήποτε νομική στιγμή η κυβέρνηση έχει την ευχαίρεια να αναστείλει τη λειτουργία μιας οργάνωσης που χρηματοδοτείται από το εξωτερικό. Τώρα εδώ οι προθέσεις είναι πολύ σημαντικές, σε αυτό θα συμφωνήσω. Όμως υπάρχει μια ενδυνάμει απειλή. Αυτοί οι περιορισμοί είναι δυνατοί και από ό,τι μπορώ να δω εγώ ουσιαστικά τίθενται σε φερμαχή. αναφέρεται και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων. Ναι, αυτό είναι σημαντικό, αλλά ο κανονισμός είναι πάρα πολύ γενικός και αόριστος. Κατά την επίσκεψή μας, εμείς ε, συναντηθήκαμε με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συνομιλήσαμε μαζί τους και μας παρουσίασαν διάφορες ανησυχίες που έχουν. Επίση, στον Παγκλαντέ συνομιλήσαμε με τον συνήγορο του πολίτη, κάποιον που μπορεί να περιγράψει κανεί ω συνήγορο. Και επίση μου είπε ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι απαραίτητη, αλλά νομίζω ότι οι μηχανισμοί στους οποίους προσφεύγει κανείς δεν θα έπρεπε να καταλήγουν ε, στην ε, αναστολή της λειτουργίας των κυβερνητικών οργανώσεων. Φυσικά μετά το 1971 υπάρχει μια αρνητική κληρονομιά. Παρ' όλα αυτά Εξακολουθώ να πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει να έχουν δικαίωμα υπεράσπισης. Στην υπεράσπιση ακόμη και όσοι κάνουν ε, εγκλήματα πολέμου. Θα ήθελα να θυμηθούμε την Ιρεμβέργη. Όλοι έχουν δικαίωμα στην υπεράσπιση. Εκτός ε, μικροφόρου, ο κ. Στάνοκ λέει ότι θέλει να απαντήσει. Ένα λεπτό κύριε Τάνοκ. Ο κύριος Βάιντεν Χόλσερ έχει ζητήσει το λόγο να... να ολοκληρώσουμε πρώτα με τον κύριο Τάνοκ ε, αυτή την διάλογο ή θέλετε πρώτα εσείς το λόγο κύριος Τάνοκ. Νομίζω υπήρχε μια παρεξήγηση. Εγώ δεν είπα ότι δεν είχε δικαίωμα υπεράσπιση σε ένας ε, εγκληματία πολέμου. Απλώς αναφέρθηκα ε, στο ότι πολύ ακριβοί δικηγόροι από το Ηνωμένο Βασίλειο χρηματοδοτούνται ε, μέσω φιλανθρωπιών με χρήματα που έρχονται από τι χώρε του κόλπου και αυτά τα χρήματα πηγαίνουν από τι χώρες του κόλπου στο Μπαγκλαντέ, σε λαφιστικές οργανώσει, ε, και πάνε να χρηματοδοτήσουν κάποιες οργανώσεις που συνδέονται με τον Τζαμάτ. Δηλαδή δεν ε, θέλω να παρεμποντιστεί η διαδικασία, των, ε, η λειτουργία των μη κυβερνητικών οργανώσεων, απλά ανέφερα ότι πολλά χρήματα μπαίνουν από εκεί και υπάρχει ριζοσπαστικοποίηση των οργανώσεων όπως ε, συμβαίνει και στη Σαουδική Αραβία, στο Κουβέιτ κτλ. Πρόκειται για μια νέα νομοθεσία που έχει ληφθεί προληπτικά. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με τη Ρωσία και το 90% του πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι στον Μπαγκλατές, όμως το κράτος έχει κοσμικό χαρακτήρα και πρέπει να προστατεύσουμε τον κοσμικό χαρακτήρα του Μπαγκλατές ως δημοκρατία. Εγώ νομίζω ότι είναι σαφή η θέση του καθένα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ο κύριο Βάιντεν Χόλτσερ, συμφωνώ απολύτω. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικός εταίρος το Μπαγκλαντέ. Θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο και υπόδειγμα προ ανάπτυξη. Είναι μια χώρα που έχει βεβαίως μεγάλη μουσουλμανική ε, πλειονότητα και μια τέτοια χώρα καταφέρνει να έχει κοσμική εξέλιξη ως κράτος. Είναι πολύ σημαντικό να αποτελέσει και παράδειγμα προς από άλλες χώρες με μουσουλμανικό πληθυσμό. Λίγες είναι οι χώρες, τα κράτη που θα μπορούσαν ε, να ε, τραβήξουν τόσο πολύ ε, μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά αυτή η νομοθεσία για τις ξένες ε, δωρεές ή συνεισφορές ε, του Foreign Donations είναι κάτι που απασχολεί πολύ και τους δικούς μας τέρους εκεί γιατί μαζί με τα ξερά κινδυνεύουν να καούν και τα χλωρά και να κατασταλούν κάποιες μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Δηλαδή υπάρχει ένα επιχείρημα και ένα αντεπιχείρημα ε, ξέρω ποια είναι η πρόθεση, ε, αλλά κινδυνεύει να έχει και άλλες συνέπειες. Και με χώρες όπως το Βαγνατές ε, ε, ε, πρέπει να συνάψουμε μια εταιρική σχέση στρατηγική για την ασφάλεια, όπως και με άλλες χώρες της περιοχής. και να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανησυχίες που αναφέρετε, αλλά μην αφορά αυτό όλες τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αν θέλετε μπορούμε και διμερώς να το συζητήσουμε, να σας εξηγήσω. Επί της ουσίας συμφωνούμε. Το ζήτημα είναι με ποιον συνεργάζεσαι και με ποιες ομάδες εκεί. Φυσικά θα πρέπει με μετριοπαθείς ε, ομάδες και μουσουλμανικές να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την κατάσταση και να αποτρέψουμε να συμβούν εξελίξεις τύπου κάποιων άλλων αραβικών κρατών. που οι μετριοπαθείς χάνουν το παιχνίδι και επικρατούν ε, ε, σελαφιστές, ε, κτλ. Θα τα δούμε σε μισή ώρα αυτά που θα ασχοληθούμε με τη Σύρια. Ευχαριστώ. Θα δώσω μέσα το λόγο στον εκπρόσωπο τη υπηρεσίε εξωτερική δράση τον κύριο Τόμας Νίκολσον, για ε, λίγη ώρα, γιατί επεκταθήκαμε πολύ. Ασχολείται με το Μπαγκλαντέ μεταξύ άλλων ε, πολλών ε, χωρών τη Ασία. Παρακαλώ. Thank Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο. Όπω και την προσωπία, και εμείς ανησυχούμε πολύ από τις πρόσφατες εξελίξεις των Μπουγκλαντές από ε, την βία χωρίς διακρίσεις, τη στοχοθετημένη βία, τις μαζικές συλλήψεις ε, πολιτικών ηγετών και από την απροθυμία από ό,τι φαίνεται και τη δυσκολία στο να προχωρήσουμε σε ένα διάλογο, να προχωρήσουν σε ένα διάλογο τα κύρια πολιτικά κόμματα μεταξύ τους. Όλα αυτά μας προβληματίζουν, όμως άκουσα σήμερα στη ζήτηση ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί τομείς όπου πρέπει να εργαστούμε με τον Μπαγκλαντές Έχουμε πολλά κοινά συμφέροντα, έχουμε καλές σχέσεις για ό,τι φορά το εμπόριο. Αναφέρθηκε ως ε, ένα πιθανό ε, παράδειγμα, υπόδειγμα σε ό,τι αφορά τις εμπορικές πτυχές και έχουμε και κοινά ανησυχίες για το θέμα της ασφάλειας, για την κλιματική αλλαγή. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό Καλωσορίζουμε την επίσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νομίζουμε είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να έχουμε σχέση με τον Μπαγκλαντές, να έχουμε δεσμεύσει και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Κομισιόν υλοποιείται μία επίσκεψη αυτή την εβδομάδα και υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις για τη διακυβέρνηση, ανθρώπινα δικαιώματα, για την ανάπτυξη, για το εμπόριο. Έτσι λοιπόν το να παραμείνουμε δεσμευμένοι είναι σημαντικό να δούμε ποιες είναι οι κοινέ μα ανησυχίε, αλλά φυσικά πρέπει να βρούμε και τις ευκαιρίες να εκφράσουμε το τι μας προβληματίζει και τι μας ανησυχεί. Έτσι, λοιπόν, νομίζω ότι πρόκειται για ένα τομέα τον οποίο θα είμαστε σε επαφή τους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ κύριε Νίκολσον. Τώρα θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους ε, της πρεσβείας. Έχει προσκληθεί η πρέσβυρα, όπως πάντα. Ε, αυτό κάνουμε όταν συζητάμε κάποια τρίτη χώρα βρίσκεται η πρεσβυρά στη Γενέβη για μια συνάντηση που γίνεται αυτές τις μέρες. Η κυρία Παρβίν θα εκπροσωπήσει την πρέσβυρα. Αν θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Και θα ήθελα να μας πείτε και ποια θα είναι η θέση του Μπαγκλαντέ σε σχέση με τη συνάντηση CDAU. Για την Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΙΕ. Ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Εκ μέρους της Πρεσβείας θέλω να ενημερώσω την υποεπιτροπή σας ότι η κυβέρνηση των Μπαγκλατές ε, ε, ευχαρίστως ε, προσφέρει τη βοήθεια στους βουλευτές από τις 16 20 Φεβρουαρίου στην επίσκεψη που υλοποίησαν. Θέλουμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας αξιόπιστος εταίρος για την ανάπτυξη για τον Μπαγκλατές και πάλι θέλω να δράξω την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας στον Μπαγκλατές, για την οικονομική οικονομική πρόοδο και επίσης σας ευχαριστούμε που το προσφέρετε ως ε, υπόδειγμα για την ε, κοσμική δημοκρατία και τη χειραφέτηση των γυναικών. Επίσης ε, θέλουμε να αναφερθούμε στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκό, Κοινοβούλιο, που θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρσι το Σεπτέμβριο και το Νοέμβριο. Και ε, αναφέρεται στη σημερινή πολιτική κατάσταση στον Μπαγκλαντές. Ε, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ε, έχουμε τρομοκρατικές δραστηριότητες από το Τζαμάτ και ολοφονούνται αυτό οι άνθρωποι με βόμβες και άλλα κτηνόδη μέσα. Όμως ο λαός του Μπαγκλαντές έχει έχει ε, ξεκινήσει ένα μπλοκάρισμα, συνεχίζει την κανονική του ζωή, ε, οι διοκτικές αρχές κάνουν τα δυνατά τους για να προστατεύσουν τη ζωή και την ιδιοκτησία των ανθρώπων. Όπως τα γνωρίζετε Πρόεδρε, κατόπιν τη υιοθέτηση του Συμφώνου Αηφορία έκανε τον Μπαγκλαντέ πολλά βήματα για να προωθήσει την ασφάλεια των εργαζομένων και κυρίως ε, στον ε, τομέα ε, RMD. Έχουμε την βελτίωση των συνθήκων εργασίας, των κτηρίων. Σε μία πρόσφατη συνεδρίαση στις 20 Οκτωβρίου εδώ στις Βρυξέλλες παρουσιάστηκαν οι αλλαγές και τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα από τα ενδιαφερόμενα μέρη όταν ε, έγινε επίσκεψη στο εργοστάσιο στην ΤΑΚΑ, ε, οι επισκέπτες έκαναν επιθεωρήσεις ε, και συμμετείχαν σε διαβουλεύσεις. Θα ήθελα να σας πω ότι όπως πάντα θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεχή μας δέσμευση και σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη του εκδημοκρατισμού. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι προς το μηδέν συμφέρον μας. Σας ευχαριστώ. Gracias. το eh, bueno, ε, Μακρηγορήσαμε λίγο, κράτησε περισσότερο από ό,τι είχαμε προβλέψει η συζήτηση. Πάντως ήταν ενδιαφέρουσα και ευχαριστώ του βουλευτέ που πήγαν στον Μπαγκλαντές για τι προσπάθειε που κατέβαλαν και ευχαριστώ εκείνου που του συνόδευσαν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να διατηρήσετε αυτέ τι επαφέ τους επόμενους μήνες με τον Παγκλαντές και να μας ενημερώνετε για τις εξελίξεις και τα τεκτενόμενα και φυσικά και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Δράσης να παραμείνετε σε επαφή και κατά κάποιο τρόπο να είστε οι πρέσβεις της δικής μας Επιτροπής για τον Παγκλαντές. Έτσι, για να μας ενημερώνετε και να μας θέλετε πάντα ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Τώρα κανονικά θα πρέπει να περάσουμε στην ανάλυση της εκθέσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τεχνολογία ο αντίκτυπο των συστημάτων παρίσπιση και παρακολούθησης τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτε χώρε. Τι έγινε? Θα δώσουμε μέσα το λόγο στην κυρία Σχάκε όταν αποχωρήσουν όσοι θέλουν να το πράξουν. les recuerdo que empezamos... Θυμίζω ότι 21 Ιανουαρίου αρχίσαμε με κοινή ακρόαση ε, με την Επιτροπή Ίντα αυτό το θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σχάκε για την ε, εκπόνηση της έκθεσης αυτής, την οποία πολύ καλά γνωρίζει. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 23η Μαρτίου το μεσημέρι και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα της δώσω το λόγο για να μας παρουσιάσει την έκθεσή της. Thank you very much, Madam Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ε, ότι είναι σαφές η τεχνολογία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και οι μαζικές ε, τεχνολογίες παρήσπιση και παρακολούθησης είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αυτή τη βδομάδα ε, μάθαμε ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου και των ε, Ηνωμένων Πολιτειών ε, είχαν ε, χακάρει τις υπηρεσίες της εταιρείας Δαμάτου που παράγει τις κάρτες σε τσίπ για τα κινητά τηλέφωνα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι υπονομεύει παγκοσμίως τα δικαιώματα των ανθρώπων και είναι εξαιρετικά οδυνηρό τέτοια παρακολούθηση, τέτοιο φακέλωμα, ιδιαίτερα αφορά ε, bloggers, δημοσιογράφους, ε, αντιφρονούντες, αντικαθεστατικούς και ε, όσους δεν συμφωνούν, εν πάση περιπτώσει. Έχει και μια ψυχή ασφαλείας που δεν μας απασχολεί ε, σήμερα, δεν είναι το παρόντος, αλλά αξίζει να το συζητήσουμε γενικότερα. Τι χρειάζεται πηγόντως να ηγηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρξει ε, νέα ε, ρύθμιση, έξυπνη, σωστή, να δώσουμε νέα σάρκα και οστά στις εμελιώδεις ελευθερίες, αρχές, τώρα που έχουμε τέτοια επαναστατική τεχνολογία. Η έκθεσή μου λοιπόν προτείνει κάποια βήματα, τα σκιαγραφή. Ήταν πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρουσα η ακρόαση που κάναμε με την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που ακούσαμε ε, ε, τον περασμένο μήνα πολλούς εμπειρογνώμονες. Οι νέες τεχνολογίες ε, προσφέρουν νέες δυνατότητες για την ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεστε, του συνέρχεστε, ε, μπορούν να βοηθήσουν για τη διαφάνεια και για την ε, λογοδοσία. Ε, όλο και περισσότερο τεχνολογικά συστήματα όμως χρησιμοποιούνται για την καταστολή. Ακούστηκε η μαζική παρακολούθηση και είναι απείρως δυσανάλογα αυτά που συμβαίνουν σε σχέση με τον επιθυμητό σκοπό, hacking, jamming, τα παράσιτα, οι υποκλοπές, οι ε, παγιδεύσεις κτλ. έχουν τεράστιες ε, επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να δούμε και τις τεχνολογικές ε, ρυθμίσει τα χαρακτηριστικά και το πλαίσιο στο οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτά είναι βασικά στοιχεία. Χρειαζόμαστε ε, πολιτική ηγεσία που να ανατρέψει, να αποκρούσει αυτό το επιχείρημα ότι η εθνική ασφάλεια μπορεί να δικαιολογεί τα πάντα. Η υπονόμευση των ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ηγηθεί θα πρέπει να δώσει εκείνη το καλό παράδειγμα και να εντάξει αυτό το είδος της θεώρησης παντού στα ανθρώπινα δικαιώματα, προγράμματα ανάπτυξης, ε, ακόμα και σε συνομιλίες ενταξιακές. Θα πρέπει να βοηθήσουμε ενεργητικά για να δημιουργηθούν και να διαδιδοθούν ε, εργαλεία, μέσα και γνώση για να μπορούν οι άνθρωποι να αυτοαμήνονται. Ε, έχει σημασία να διδάξουμε τον κόσμο, να το διαπαιδαγωγήσουμε για το πώς μπορεί να χρησιμοποιεί και με ασφάλεια να προστατεύει την ιδιωτική του σφαίρα για να μην παραβιάζονται ούτε τα έγγραφα ούτε οι αρχές και οι δικαιώματα. Θα πρέπει να συνεργαστούμε και με δικαστήρια και με ειδικού ε, για στα δικαστικά θέματα, εμπειρογνώμονε, για να δούμε πώ όλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται στα δικαστήρια. Δυστυχώ σήμερα δεν ηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε σε πολιτικό επίπεδο, ούτε γενικότερα. Υπάρχουν πάρα πολλέ τεχνολογίε που χρησιμοποιούνται ε, για να υπονομεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και μιλάμε εδώ πέρα για ένα κλάδο της ε, πολλών εκατομμύριων δολαρίων. Χρειάζεται έξυπνη αντιμετώπιση, ε, συνολική. Δεν μπορεί να είναι ε, διακρατική υπόθεση μεταξύ δύο κυβερνήσεων κάθε φορά, διμερές θέμα. Ε, επίσης, η εξαγωγή των τεχνολογιών αυτών, η hacking, υποκλοπές και μαζική παρακολούθηση χρειαζόμαστε και ε, μελέτες αντικτύπουν και να βάλουμε και ερωτηματικά ε, στα πρότυπα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την νόμιμη δυνατότητα υποκλοπής που ζητούν ε, στα δίκτυα των τηλεπικοινωνιών. Αλλά όταν χρησιμοποιούνται παράνομα αυτά είναι τελείως διαφορετικές οι επιπτώσεις. Τι σημαίνει αυτό. Όταν υπάρχει ένα τεχνικό παραθυράκι που μπορεί να ανοίξει στην Ευρώπη μόνο μετά από ένταλμα η εντολή ε, δικαστική, ε, εντάξει, αλλά τι γίνεται όταν το κάνουν σε τρίτες χώρες αυτό, μυστικές υπηρεσίες, διοκτικές αρχές, αστυνομία και κυβερνήσεις, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Ε, θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ευάλωτα σημεία στα λογισμικά μας που μπορούν να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης και κατάχρησης. Επίση, να δούμε τι γίνεται από την ε, επιχείρηση καταστολή των κυβερνήσεων που αφορούν και λογοκρισία και άλλη περιστολή ελευθεριών και έχουν και το μανδύα ε, της νομιμοποίησης με το επιχείρημα λέει, της ε, ε ασφάλειας ή τα διεθνή φόρα για το ίντερνετ, IGF, ITU και άλλα. Και εκεί χρειάζεται να αναλάβει τα ενία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, προχωρούμε και εξετάζουμε τα διάφορα ε, μέσα που μπορούμε να αναπτύξουμε. Θα πρέπει να, να φροντίσουμε να μην ε, εμποδίσουμε ε, την νόμιμη χρήση, ούτε να υπονομεύσουμε την έρευνα που γίνεται, που είναι πολύτιμη σε αυτές τις τεχνολογίες. Μπορούμε να βρούμε όμως μια σωστή ισορροπία και βασιζόμενη στην εμπειρία της ακρόασης Έχω βάλει το σχέδιο έκθεση και στη δημόσια διαβούλευση, στο διαδίκτυο. Η κοινωνία των πολιτών να τα δουν οι πυρογνώμονε, οι hackers, οι ειδικοί να μα πούν τη γνώμη του για να μα προτείνουν πώ να καταρτήσουμε αυτή την νομοθεσία και προσβλέπω στη συνεργασία με τους συναδέλφους για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η έκθεση. Ε, η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι 23 Μαρτίου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σάκε. Νομίζω ότι η τοποθέτησή σας ήταν εξαιρετική. Ε, καταλάβαμε πολύ καλά ως Επιτροπή τι πρέπει να προωθήσουμε και γιατί πρέπει να ενδιαφερθούμε ακριβώς. Έχουμε σκιώδεις εισηγητές που θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή να πάρουν το λόγο, εάν το επιθυμούν. Για να δω. Η κυρία... Α, ο κύριος Γιώσεφ Βάιντενχόρσεφ. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο και ο κύριος Τζι. Γκρζίπ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σήμερα ε, αντικαθιστώ εδώ και γι' αυτό παίρνω άλλωστε το λόγο την κυρία Γκότλιφ, σκιώδη συγγήτρια, για το θέμα αυτό, διότι δεν μπόρεσε να ε, είναι εδώ για προσωπικούς λόγους και γι' αυτό μου ζήτησε να σας ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της και να παρουσιάσω την άποψή της για την έκθεση που ε, ανέπτυξε η κυρία Σάκε. Είπατε ότι οι εξελίξεις στην τεχνολογία ε, της πληροφορικής και ο αντίκτυπος του στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι το πολύ σημαντικό σήμερα και πράγματι ισχύει αυτή η δήλωση και εγώ τη συμμερίζομαι. Είμαστε μάρτυρες μιας τεράστιας επανάστασης, επανάστασης της τεχνολογικής και πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή γιατί η τεχνολογία δεν χρησιμοποιείται πάντοτε για καλούς σκοπούς, για την ανάπτυξη, για την καινοτομία, αλλά χρησιμοποιείται ε, για να καταστρατηγηθούν ανθρώπινα δικαιώματα, ακτιβιστών και άλλων. Η σκιώδης λοιπόν η συγγήτρια ευχαριστεί την κυρία Σάκε η οποία συνέταξε μια περιστατωμένη και εξισορροπημένη έκθεση, η οποία είναι πολύ σημαντική, διότι η ελευθερία θα πρέπει να συμπληρώνει την ψηφιακή ασφάλεια και αντιστρόφως. Πρέπει να ενισχύσουμε τη θέση των στρατευμένων ε, υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας, να προωθήσουμε το δικαίωμα στην ιδιωτική σφαίρα, να ενισχύσουμε ε, την ελευθερία του εκφράζεστε, την ελευθερία του συνεταιρίζεστε, ε, τη συμμετοχή σε οργανώσεων και μάλιστα και σε διαδικτυακό ε, τοπίο. Και ξέρετε, όλες αυτές οι διαδικτυακές πλατφόρμες παίζουν σημαντικό ρόλο σε απολυταρχικά καθεστώτα. Εκεί όπου έχει αυξηθεί η πρόσβαση στη ψηφιακή ελευθερία, τα τελευταία χρόνια έχουμε θετικές εξελίξεις και έχει δράσει καλύτερα η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμισε πρόσφατα ε, ε, πόσο απαραίτητη είναι η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά τα μέσα. και ε, στο πεδίο των εμπορικών διαπραγματεύσεων και του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την ε, ενταξιακή πορεία οποιασδήποτε χώρας. Επομένως, θα πρέπει να εξετάσουμε και τις αρνητικές συνέπειες κάθε φορά που εισάγουμε νέες τεχνολογίες και αυτό θα πρέπει να φανεί στη διατύπωση του κειμένου. Και να έχουμε μία σωστή ισορροπία για να αποφύγουμε συνέπειες που δεν επιθυμούμε. Οι απαγορεύσεις π.χ. αυτές δεν πρέπει να έχουν να κάνουν με την έρευνα στις νέες τεχνολογίες ή για τις τεχνολογίες που είναι απαραίτητες στην ανάπτυξη των χωρών. Ωστόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο έχει ηγετικό ρόλο και στον τομέα της ψηφιακής ελευθερίας και ασφάλειας και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γι' αυτό πρέπει να εκπέμψουμε το χειρό μήνυμα ότι δεν μπορεί κανείς να ε, χρησιμοποιεί την τεχνολογία της πληροφορικής για να παρεμποδίσει την άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα δικαιώματα όσων επιχειρούν, τα δικαιώματα όσων είναι ακτιβιστές και το καθεξής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Βάιντεν Χόλσερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Η έκθεση είναι πάρα πολύ εκτενής. Οι συζητήσεις ε, της περασμένης ακρόασης έχουν ε, συμπεριληφθεί πάρα πολύ καλά στην έκθεση. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη και ε, τα επικεντρώνει όλα πάρα πολύ καλά. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα παραλληλισμό ε, με τα όσα συμβαίνουν στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για μια ψηφιακή habeas κόρπους. Νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε τις δυνατότητες αυτοπροστασίας του ατόμου για την κρυπτογράφηση και θα ε, ε, πρέπει όλοι να ε, αντικρούσουμε όλες τις απόπειρες που γίνονται παραβίασης. Ξέρουμε ότι είναι ένας πολύ μεγάλος κλάδος της οικονομίας αυτό. Για αυτούς τους λόγους δεν θα πρέπει να είναι οι ρυθμίσει αυτές εθελούσιε, αλλά να ζητούμε και δεσμευτικέ. Συμφωνώ με την εισηγήτηρια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει το ρόλο που της αναλογεί, που είναι πρωταγωνιστικός και ηγετικός και πρέπει και παγκοσμίω κάπως να φανούμε, να προβληθούμε. Και αν δεν το κάνουμε εδώ, πού θα το κάνουμε. Ευχαριστώ. Sí, muchas gracias, señor Panzeri. Ευχαριστώ, κύριος Παντζέρη. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα στη βάση της συζήτηση που γίνεται και έχει δηλοποιηθεί, πέρα από την αξιολόγηση των θετικών ή αρνητικών συνοπιών ε, της ε, τεχνολογικής κινητομίας ε, στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμείς να ήμασταν σε θέση, στα πλαίσια της έκθεσης αυτής, να εισαγάγουμε την έννοια της δημοκρατίας, της τεχνολογικής δημοκρατίας. Πρέπει να ορίσουμε νέα πρότυπα. Βεβαίω, αυτό είναι μια πολύ δύσκολη διαδρομή, μια πολύ δύσκολη διαδικασία, γιατί βρισκόμαστε ενώπιον μιας ε, καινοτομίας. Ε, αν και έχει επέλθει εδώ και καιρό, αλλά εμεί θα έπρεπε να εργαστούμε επί νέων κριτηρίων που να ορίζουν την έννοια τη τεχνολογική δημοκρατία, γιατί είναι ο μόνο τρόπο για να διαχειριστούμε καλύτερα αυτή τη διαδικασία και τις επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι λοιπόν, εγώ θα ήθελα να αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε επί αυτού του θέματο. Αυτό ζητάω. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν η κυρία Σάκε θέλει να απαντήσει, να πει κάτι. Συγγνώμη κυρία Σαρτζεντίνη, δεν μου πέρασαν το όνομά σας, δεν μου το διαβίβασαν, αλλά όποτε θέλετε έχετε το λόγο φυσικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ήθελα να συμπληρώσω το εξή. Νομίζω ότι είναι Πολύ καλό το χρονικό διάστημα που έρχεται η έκθεση της ε, κυρία Σάκε και ε, νομίζω ότι ε, φυσικά πάντοτε η μαζική παρακολούθηση είναι δυσανάλογη. Συμφωνώ με αυτό και θα ήθελα να επενθυμίσω ότι πέρσι ο Σνόντεν ήταν ο δεύτερος, δεύτερο, ήρθε δεύτερος για το βραβείο Ζαχάροφ και υπήρχε υποστήριξη από όλες τις ομάδες. Και επίσης, μετά την επίθεση στο Σαρλί Εμπτό, ξέρουμε ότι η συζήτηση περί ασφάλειας και ερευνά έχει τεθεί επιτάπητο. Επομένως, εγώ ανησυχώ ότι δεν θετούμε το κατάλληλο παράδειγμα εδώ, δεν δίνουμε το κατάλληλο παράδειγμα. Θέλω να υπενθυμίσω τη συζήτηση που έλαβε χώρα στη Ρήγα στο Συμβουλίο των Υπουργών στα τέλη Ιανουαρίου, στο Συμβουλίο Υπουργών Δικαιοσύνη, όπου ο συντονιστής εξήγησε στους υπουργούς μας ότι από τις αποκαλύψεις του Σνόντεν και μετά υπάρχει μία τάση οι άνθρωποι να ε, προβαίνουν σε αποκεντρωμένη προστασία και κρυπτογράφηση και είπε ότι αυτό είναι επικίνδυνο γιατί δεν θα επέτρεπε στις εθνικές αρχές να ερευνήσουν, καθώς οι άνθρωποι έχουν προστατευτεί τόσο καλά και πρότεινε η Κομισιόν να υποχρεώσει τις ε, εταιρείες τηλεπικοινωνιών ε, και διαδικτύου να δίνουν πρόσβαση χωρίς όρους σε αυτούς τους κώδικες. Τώρα αν κάνουμε αυτό, αν στην Ευρώπη προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τη μεμονωμένη ασφάλεια των ανθρώπων στο διαδίκτυο, τι θα σημαίνει αυτό για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εξωτερικό. να δώσουμε το σωστό παράδειγμα είναι ζωτικό, είναι θεμελιώδου σημασίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξαγωγή της νομοθεσίας ε, και ε, υλικού, λογισμικού σε καθεστώτα καταπιαστικά Πώς είμαστε σίγουροι ότι θα εμποδίσουμε τέτοιες εξαγωγές. Πολλές φορές το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την καταστολή ενός προσώπου είναι το ίδιο λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιον άνθρωπο για να αυτοπροστατευτεί. Το λογισμικό δεν είναι κάτι που μπορούμε να το επιλέξουμε. Αν ε, παραδείγματος χάρη απαγορεύσουμε την εξαγωγή όπλων ε, ενός ΤΑΝ και αυτό είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Όμως ε, για το software μιλάμε εδώ για κωδικό ότι αποκαλύπτεται ο κωδικός. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες ε, δεν κερδίζουν χρήματα πολλώντας προϊόντα σε καταπιεστικά καθεστώτα που οδηγούν σε περισσότερη καταστολή αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ε, οι υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, να μπορούν να κάνουν ε, τη δουλειά τους επιγραμμικά και να μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό του με αυτό το λογισμικό. Επίσης, νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε το θέμα της ε, χειραφέτησης, της ενδυνάμωσης των ανθρώπων αυτών που περισπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό είναι μέρος ε, των προτάσεων που είναι επιτάπητος και από την κυρία Σάκη και θα έπρεπε να διερευνήσουμε και τις δυνατότητες, πώς αυτό θα το πλαισιώσουμε έτσι ώστε να μην είναι αδύνατο το ευρωπαϊκό λογισμικό να χρησιμοποιείται από τις περισπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σακεντίνη. Κυρία Σάκη για να ολοκληρώσει. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σα και βλέπω να υπάρχει τέτοιο περιθώριο, υπάρχει δυνατότητα να προσθέσουμε ε, και άλλα στοιχεία στην έκθεση αυτή. Μας περιορίζει ο περιορισμένος αριθμός χαρακτήρων βέβαια. Τώρα για να απαντήσω στα θέματα που έθεσε η κυρία Σαρτζεντίνη δεν είναι εύκολο ταυτόχρονα. Όταν ε, εξετάζουμε τι μπορεί να γίνει στο πλαίσιο των εμπορικών μέτρων, εντοπίζοντας κάτι ως δυτή χρήση δεν έχει γίνει ε, για πρώτη φορά αποτελεσματικά. το χάρη ένα μαχαίρι μπορεί να κόψει κάποιο το ψωμί αλλά μπορεί και να σκοτώσει κάποιον. Έτσι λοιπόν εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το πλαίσιο και αν δούμε τον κανονισμό περί εξαγωγών και εγώ ως μέλος της Επιτροπής Εμπορίου έχω εργαστεί στο θέμα αυτό Άντε αρχίσαμε να μιλάμε για οικονομικές ε, συμφωνίες που γίνονται με εταιρείε που έχουν έδρα στην Ευρώπη και κυβερνήσεις τρίτων χωρών, διοκτικές αρχές, επιχειρήσεις δημόσιες όπως οι εταιρείε τηλεπικοινωνιών, τότε αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε την αγορά των συστημάτων αυτών και θα ήθελα να σας παροτρύνω όλους ε, να δείτε ε, και το κατάλογο, ε, διεθνό κατάλογο, όπου υπάρχουν κάποια από τα υλικά που τη σε εμπορία από αυτές τις εταιρείες και πολύ συχνά δεν είναι δυνατόν να υπάρχει πολλαπλή ερμηνεία για το στόχο χρησιμοποίησης αυτών των συστημάτων. Επίσης, ε, πρέπει να δούμε και πώς μοιραζόμαστε του συμβούλους, ε, τις συμβάσεις υπηρεσιών, την ανάπτυξη στο δεύτερο των χωρών. Ξεκάθαρα βλέπουμε ότι αυτά τα συστήματα δεν χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένους φορείς και ανθρώπους, είναι για μία και μόνη χρήση. Και πιστεύω ότι για την επιβολή του νόμου ή αν δούμε τις απαιτήσει ε, να έχουν άδεια οι εταιρείε ε, πριν εξαγάγουν αυτά τα συστήματα, ε, να έχουμε τα μέσα να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ ενός ερευνητή, ο οποίος στο πλαίσιο της ερευνά του θέλει να έχει πρόσβαση σε αυτό το λογισμικό και άλλων τεχνολογιών και των πρωταγωνιστών στην αγορά που προσπαθούν να πουλήσουν. Και πολύ συχνά έχουν ε, δηλώσει ότι σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχεδόν ε, καμία νομοθεσία και καμία απέτηση αδειοδότησης. Επειδή υπάρχει έλλειψη διαφάνεια στο ποια συστήματα είναι αντικειμενοπορίες και το ποιε είναι οι επιπτώσει, επιτρέπουμε σε μία ήδη σκοτεινή αγορά εταιριών, μιλάμε για εταιρείε που μάλλον δεν έχουμε ακούσει ποτέ τα ονόματά τους, να κάνουν πραγματικά δρόμικες δουλειές. Έτσι λοιπόν, ε, εγώ τονίζω εδώ τι οικονομικέ συναλλαγές, να δούμε τι απαιτήσει αδειοδότηση. Αν το κάνουμε αυτό, θα μπορούμε να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ του θεμητού σκοπού, δηλαδή να χρησιμοποιούνται από ερευνητέ, από ερευνητέ ανθρώπινων δικαιωμάτων κτλ. και του μη νόμιμου σκοπού, δηλαδή από ανθρώπου που θέλουν να καταστήλουν. Και εδώ ε, πρέπει να υπάρχει ένα περιορισμό γιατί αυτέ τι τεχνολογίε μπορούν να πολυθούν και σε εγκληματικέ οργανώσει και να έχουμε έτσι τεράστιε αρνητικέ επιπτώσει ε, επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια ευρεία προσέγγιση, να λάβουμε υπόψη και το θέμα της ασφάλειας ε, και της στρατηγικής. Έτσι λοιπόν, για μένα εδώ υπάρχουν πάρα πολλές σημαντικές πτυχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ελπίζω στον επόμενο μήνα μέχρι την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τους εμπειρογνώμονες και να εκπονήσουμε κείμενα διατυπώσεις έτσι ώστε να στοχεύσουμε σε αυτούς που πρέπει να στοχεύσουμε και να μην έχουμε ανεπιθυμητές συνέπειες. Πρέπει τουλάχιστον να κάνουμε μια αρχή, γιατί τώρα νομίζω ότι είναι απαράδεκτο το status quo. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σχάκε. Καλό όλους τους συναδέλφους να συνεργαστούν με την εισηγήτρια στην εκπόνηση τη έκθεσης με τις τροπολογίες. Περνάμε λοιπόν τώρα στην ακρόασή μας σχετικά με την ελευθερία θρησκείας, υπεπιθύσεων ή συνείδησης όπως θέλετε να την ονομάσετε για τους χριστιανούς και άλλες σκεφτικές μειονότητες στη Μέση Ανατολή. Θελήσαμε να προετοιμάσουμε αυτή την ακρόαση, να τη διοργανώσουμε, γιατί θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό ε, να αναλύσουμε την κατάσταση εκεί, της έλλειψης ουσιαστικά ελευθερίας, ε, θρησκείας ή συνείδησης σε πολλές χώρες μέσα Ανατολής. Βέβαια διαφέρουν οι χώρες και οι καταστάσεις, αλλά σαφέστατα διώκονται οι μειονότητες και ιδιαίτερα οι χριστιανοί. Ήδη το 2013 το Συμβούλιο ενέκρινε τις ε, ε, κατευθείας γραμμές τους προσανατολισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελευθερία συνείδησης και θρησκείας. Αυτή είναι παλιά ε, φιλοδοξία και προσδοκία της ανθρωπότητας, αλλά εξακολουθεί να απουσιάζει από πολλές χώρες του κόσμου. Ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή η κατάσταση είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Πέρυσι ε, ε, ε, η τρομοκρατική ομάδα Ντάες ανέλαβε την ευθύνη για την εκτέλεση 21 σκοπτών Αιγυπτίων, χριστιανών και σε βίντεο μάλιστα. Και εμείς ζητήσαμε στην Σαουδική Αραβία να αφαιθεί ελεύθερος ο Ραϊφ που είναι ε, δημοσιογράφος και blogger και έχει δημιουργήσει έναν ιστότοπο για τις συζητήσεις ε, με θέματα θρησκείας και ε, ελευθερίας και αυτό το θεώρησε βλασφημία το καθεστώς και το καταδίκασαν σε 10 χρόνια φυλάκιση και σε χίλιους σε χίλια ραπίσματα. Επανειλημμένα έχουμε ε, καταδικάσει αυτά τα φαινόμενα της παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς ε, και τις συσκευτικέ ελευθερίες. Μαζί με την αντιπροσωπεία για το ΜΑΣΡΕΚ, ε, που προεδρεύει η κυρία Μαρίσα Ματίας και θα μιλήσει στη συνέχεια, διοργανώνουμε τη Μαρούσα Ακρόαση. Έχουμε ενώπιόν μας ανθρώπους πάρα πολύ ε, δεσμευμένους και στρατευμένους σε αυτή την υπόθεση της προστασίας της ε, ε, ελευθερίας και θα πρέπει να παραμείνουν ελεύθερες οι συνειδήσεις εκεί. Ο Πάτερ Νάμα Σαμόρ που είναι η Σουήτης, από ένα καταφύγιο Σουητών στην Συρία, ο κύριος Ντανιέλ Χόφμαν από το Middle για να μας πει γενικά πώς έχει η κατάσταση είναι ο κύριος Βουίλιαμ Σπένσερ, εκτελεστικός διευθυντής ε, του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η κυρία Άλισον Σμιθ, διευθυντήρια ε, του προγράμματος Διεθνούς Πυρικής Δικαιοσύνης «Καμία ειρήνη χωρίς ε, δικαιοσύνη» και την κυρία Αστέρ Κάτεμπερκ ε, έχουμε και τον πατέρα Μουράντ Αμπού Σεϊφ, ε, διευθυντή του προγράμματος των Ιησουητών που ε, εργάζεται στο Χαλέπι και έχει τρομερή ίδια εμπειρία και γνώση. Δεν θέλω να επεκταθώ. Εγώ θέλω να δώσω πρώτα το λόγο στον πατέρα Ναουρα Σαμούρ για 15 λεπτά το πολύ. είναι τιμή και χαρά για μένα που βρίσκομαι μαζί σας εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή. Ξέρετε, είναι περίπλοκο και ε, δύσκολο Αυτά μπορώ να πω για την κατάσταση στη Συρία σήμερα μετά από τέσσερα χρόνια τοπικού πολέμου ανελέητου με τεράστιες και τραγικές συνέπειες σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι πολλές και διαφορετικές, οι πρωταγωνιστές των συγκρούσεων είναι πολλοί και διαφορετικοί, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανείς ελεύθερα στη χώρα, δεν μπορεί να, έχει, να βρει εθνικό ή διεθνή τύπο που να απεικονίζει την πραγματικότητα και την καθημερινότητα των Σύριων πολιτών με αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο. Και για όλους αυτούς τους λόγους το να καταλάβει κανείς την πραγματικότητα στη Συρία και να την εξηγήσει είναι σχεδόν αδύνατη αποστολή. Ε, οι γνώσεις που έχουμε αποκτήσει και οι εμπειρίες που έχουμε βιώσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τις οποίες συνειδητοποιούμε ε, εκ των υστέρων, ουσιαστικά αποτελούν ένα μικρό κομματάκι μόνο της πραγματικά, πραγματικής αληθινής καθημερινής ζωής που ζουν οι, σήμερ, οι Σύριοι σήμερα. Και γι' αυτό θα ήθελα να επαναλάβω πόσο περίπλοκη και ε, μπερδεμένη είναι η κατάσταση. Θα ήθελα να προσπαθήσω να εξηγήσω και ε, σε άλλους αλλά και στον εαυτό μου ορασμένα πράγματα που μας έχουν επιβληθεί ε, στη Συρία. Και ε, χάρη σε άλλους ε, ε, χριστιανούς και μουσουλμάνους προσπάθησα σαν χριστιανός που είμαι και προσπαθώ πάντοτε να απαντήσω με δίκαιο τρόπο σε αυτό το ερώτημα. Πώς μπορεί κανείς να αντέξει, δηλαδή πώς να διατηρήσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε απάνθρωπες συνθήκες, πώς μπορεί να κάνει το καλό ξεκινώντας από την αδυναμία, την έλλειψη πόρων και την εγκύτητα του θανάτου. Εγώ δεν μπορώ βεβαίως να δώσω την χριστιανική απάντηση. Η, απάντηση που θα δώσω είναι η δική μου. Μία δυνατή απάντηση μεταξύ πολλών άλλων. Τα γεγονότα στη Συρία ξεκίνησαν την άνοιξη του 2011 και μετά από την περίοδο των διαδηλώσεων στην αρχή σιγά σιγά η χώρα γλίστρησε σε αυτή την ομή βία. Είναι μια κρίση βεβαίως παγκόσμια, συνολική. Ε, είναι μια κρίση που αγγίζει το σύνολο της χώρας σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Και παρά ε, ε, υποτίθεται την ε, βιτρίνα της ε, σταθερότητας η οποία είναι μια ψευδέστηση και παρά την ευημερία η οποία κατ' επίφαση μόνο μπορεί να ονομαστεί ευημερία η Συρία δεν είχε τις απαραίτητες δομές για να εξυγχρονίσει το κράτος και να ε, είναι βιώσιμη και γι' αυτό είμαστε εν μέσω κρίσης και θα ήθελα να προσπαθήσω να δώσω την εικόνα του τι εστί πραγματικότητα Συρία τι είναι αυτή η χώρα και τα χρώματα με τα οποία θα την περιγράψω είναι αρκετά ε, μελανά χρώματα, γιατί σήμερα η κρίση έχει αλλάξει τα πάντα. Ο φόβος, η ανησυχία, η ασφάλεια. η οδύνη είναι η μοίρα όλων μας. Κανένας Σύριος ούτε φανταζόταν ούτε είχε επιθυμήσει ποτέ η Συρία να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ποτέ δεν είχαμε φανταστεί ούτε επιθυμήσει να ζήσουμε μια τόσο τραγική ε, κατάσταση. Ε, δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο στη Συρία που να είναι ήσυχο, που να μην υπάρχουν βιαιότητες και ε, φρικαλαιότητες. Σήμερα στη Συρία το μόνο που υπάρχουν είναι εκτιμήσεις, δεν έχουμε επίσημες στατιστικές και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η θάνατοι είναι άνω των 210.000, 15.000 με... μεταξύ των οποίων είναι παιδιά, ένα εκατομμύριο ή τραυματίες και δυστυχώς τα νούμερα αυτά δεν μου φαίνονται καθόλου αντιπωσιακά. Πιστεύω ότι είναι είναι μάλλον πραγματικά, ρεαλιστικά και δεν αναφέρομαι καν ε, στους ε, ε, εξαφανισμένους, στους αγνοούμενους, όσοι έχουν, είναι υποκράτηση, έχουν απαχθεί και ούτω, καθεξή, ούτω καθεξής. Γίνεται λόγος για 7,6 εκατομμύρια ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί, έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους χωρίς τίποτα να πάρουν μαζί τους, εκτός από τα ρούχα τους, για να ξεφύγουν από αυτή την αυθαίρετη βία χρειάζονται τα πάντα είναι άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί επανειλημμένως, έρχονται σε ένα μέρος που ήταν ήσυχο και μετά υπάρχει νέο κύμα βίας και αυτός ο εσωτερικός πρόσφυγας πρέπει να εγκαταλείψει και το καινούριο μέρος για να πάει σε ένα τρίτο μέρος και ούτω καθεξής. Και έχουμε και τους εκτοπισμένους που έχουν υποστεί τις συνέπειες των γεγονότων, την ανεργία και ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. 12,12 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επιγόντως ανάγκη από βοήθεια. Και έχουμε και 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους που εγκατέλειψαν οριστικά ε, τη χώρα και πήγαν στις γειτονικές χώρες. Σήμερα στη Συρία το ποσοστό εγκληματικότητας είναι εξαιρετικά υψηλό. Έχουμε απαγωγές, έχουμε λιστίες σε σκοτώνουν για χρήματα, σε απαγάγουν για λίτρα, νέα φαινόμενα στην ε, ε, κοινωνία των Σύρων. Είμαστε μάρτυρες της εξαφάνισης όλων των απαραίτητων υποδομών για τη ζωή. Μιλούμε για υποδομές μεταφορών, για νοσοκομεία, για σχολεία, δεν υπάρχει τίποτα. Ο δημόσιος τομέας είναι ανύπαρκτος οι δυνατότητές του είναι κάτω από ε, τις μισές από αυτές που είχε πριν από ε, την κρίση. Βεβαίως μιλούμε για την άνοδο του, ε, ριζ, της των θεμελιωδών, ε, των φονταμεταλιστικών ομάδων. Έχουμε το isis το Νούσρα, το Ισλαμικό μέτωπο. Όλοι αυτοί θέλουν να φτιάξουν ένα Ισλαμικό κράτος. Ίσως διαφορές έχουν μικρές μεταξύ τους, αλλά προσπαθούν να επιβληθούν σε όλη τη Συρία και σε όλη την περιοχή. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι αυτοί που κυβερνούν σήμερα υποτίθεται τις, ε, τις υποτίθεται απελευθερωμένες ζώνες. Αναρωτιέμαι, πρόκειται πράγματι για απελευθερωμένες ζώνες. Και ξέρετε, σε διεθνέ επίπεδο μιλούμε για τη στήριξη των μετριοπαθών ομάδων. Εγώ είμαι σύρος και προσπαθώ να είμαι όσο δυνατόν πιο αντικειμενικός. Υπάρχει τέτοιο πράγμα, υπάρχει μετριοπάθεια, υπάρχουν μετριοπαθείς ομάδες. Δεν λέω ότι δεν υπήρχαν, λέω σήμερα αναρωτιέμαι, υπάρχει κάποιο μετριοπαθή. Μία άλλη βεβαιότητα που με συγκλονίζει είναι το γεγονός ότι ο πόλεμος είναι αιματηρός αλλά εξαιρετικά τοπικός, στη Συρία μόνο και σε λίγα εδάφη του Ιράκ. Και οι επιπτώσεις όμως αυτού είναι διεθνείς. Επηρεάζουν όλη την περιφέρεια και επηρεάζουν και το διεθνές πολιτικό γίγνεσθε. Θα μπορούσε κανείς αυτό να το εξετάσει υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες. Πράγματι, πρόκειται για εμφύλιο πόλεμο στη Συρία. Όμως, θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι Κούρδοι είναι εναντίον των ε, ε, Τούρκων, οι Σιήτες των Σουνιτών, η Δύση εναντίον της Ανατολής και το καθεξής. Ένα άλλο σκοτεινό σημείο και θέλω να το τονίσω ως χριστιανός είναι η, η αβεβαιότητα της χριστιανικής κοινότητας. Όλοι οι Σύριοι είναι ανήσυχοι, όλοι οι πολίτες, κανείς δεν έχει το μονοπόλιο της οδύνης, όλοι υποφέρουν, είναι κάτι γενικευμένο και γενικό. Λόγω της ανόδου του ε, ριζοσπαστικού Ισλαμισμού και λόγω των τραυμάτων ε, της βίας που έχει υπάρξει στις γειτονικές χώρες, το Ιράκ, το Λίβανο κτλ, η στάση των ε, χριστιανών είναι πολύ μεγαλύτερη η ανησυχία τους από την ανησυχία άλλων πολιτών της Συρίας, άλλων θρησκευμάτων. Όλο και περισσότερο κυριαρχούν εξτρεμιστικά κινήματα που έχουν τους χριστιανούς ως πρώτο στόχο και είδαμε τις φρικτές σκηνές πριν από τρεις μέρες που εκτελήχθηκαν στη Συρία. Οι χριστιανοί λοιπόν πλήττονται όπως και οι άλλες μειονότητες ακόμα και οι ε, φιλελεύθεροι Σουνίτες, διότι ο ριζασπαστικός φονταμενταλισμός υιοθετεί μια μανιχαϊστική άποψη του κόσμου. Για αυτούς υπάρχουν μόνο όσοι κατέχουν την αλήθεια και αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά υπάρχουν όλοι όσοι δεν ανταποκρίνονται στο όραμα και στο πρόγραμμά τους και αυτοί πρέπει να καταπολεμηθούν και να εξαλειφθούν γιατί ε, βάσει αυτής της μανιχαϊστικής προσέγγισης αυτοί οι τελευταίοι ενσαρκώνουν το απόλυτο κακό. Επομένως οι χριστιανοί είναι ο αδύναμος ε, κρίκος ε, της ε, κοινωνίας και ελοχεύει ο κίνδυνος στο κεφάλι τους να πέσουν όλες αυτές οι αρνητικές συνέπειες, να βιώσουν αυτό τον φρικτό αντίκτυπο ε, πολύ πιο έντονα και ισχυρά από ό,τι οι υπόλοιποι. Και γι' αυτό οι χριστιανοί της Συρίας περνούν την πιο φρικτή δοκιμασία σήμερα. Ε, μιλούν πάντοτε για κάτι που είναι αλλού, στο εξωτερικό. Ε, είναι σπίτι τους, αλλά είναι ε, απομονωμένοι, είναι, νιώθουν ξένοι οι περισσότεροι επιθυμούν να φύγουν και μάλιστα νιώθουν αυτή την αποξένωση και τη χρονική γιατί ή ασχολούνται με το λαμπρό παρελθόν ή ελπίζουν για ένα ε, καλύτερο μέλλον. Δεν μπορούν να ζήσουν στο παρόν αυτή τη στιγμή. Δεν ζουν στο παρόν και αυτό είναι δυστυχές. Είναι πολύ κρίμα. Δυστυχώς σήμερα στη Συρία ε, ο θάνατος είναι κάτι, είναι μια κοινοτοπία πλέον, είναι μπανάλ σχεδόν θα έλεγα. Ε, μπορεί να χτυπήσει τον καθένα οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Είναι δραματική η κατάσταση. Τίθεται το ερώτημα, υπάρχει χώρος για την ελπίδα, πώς μπορεί κανείς να αντέξει σε τέτοιες απάνθρωπες συνθήκες ε, στις οποίες διαβιούμε σήμερα. Με αυτό το μελανό τοπίο λοιπόν μπορούμε ακόμα να ελπίζουμε αν θέλω να είμαι ρεαλιστής και ορθολογιστής που επιθυμώ συνήθως να είμαι θα έλεγα τότε ότι δεν υπάρχει πλέον τίποτα να κάνουμε. Απολύτως τίποτα. Ωστόσο είμαι χριστιανός, είμαι πιστός, είμαι ιερέας και δεν έχω δικαίωμα να πω κάτι τέτοιο. Εκεί όπου δεν υπάρχει πλέον τίποτα να γίνει, εκεί είναι που πρέπει όλα να ξαναγίνουν από την αρχή. Απολύτως όλα. Και γι' αυτό πρέπει να έχουμε επινοητικότητα, εφευρετικότητα για να μπορέσουμε να χαράξουμε και να ανοίξουμε δρόμους. Ως GRS ε, οι ουσίτες στη ε, Συρία, οι οι Σουίτες στη Συρία, ε, στη Δαμασκό προσπαθήσαμε να ανοίξουμε ένα δρόμο και έχουμε ιστιά έχουμε ε, ε, το σπίτι που υποδέχεται τους ανθρώπους. Σήμερα μετά από τέσσερα χρόνια σύγκρουσης, 28.000 οικογένειες βοηθούμε. Κάθε βράδυ παίρνουν το καλάθι σύντησής τους και έχει τρόφιμα, έχει ήδη ε, πρώτης ανάγκης για να μπορέσει να ζήσει μια οικογένεια κανονικά, αν και δεν ξέρω πια τι θα πει κανονικά, τι θα πει normal. Έχουμε κέντρο φροντίδας των ε, πασχόντων που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες και που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα βασικά τους φάρμακα. Και προσπαθούμε επίσης να ε, βοηθήσουμε όσους έχουν ιατρικές ανάγκες παραπέμποντας τους ενίοτε στα νοσοκομεία. Ε, τρίτο σκέλος της εργασίας μας, τα παιδιά τα παιδιά τα οποία έχουν υποστεί τεράστια τραύματα. Μιλούμε για χιλιάδες παιδιά. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτά. Προσπαθούμε να ανοίξουμε τα κέντρα μας και βοηθούμε σχεδόν 6.000 παιδιά. Ε, προσφέρουμε στήριξη ψυχοκοινωνική και προσπαθούμε να καλυφθούν τα εκπαιδευτικά τους κενά για να μπορέσουν να έχουν ελπίδα για ένα μέλλον. Προσπαθούμε να ε, έρθουμε σε επικοινωνία με τις οικογένειές τους, να οργανώσουμε δραστηριότητες. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε δεν απευθύνονται μόνο σε χριστιανικές οικογένειες. Αντιθέτως, όλοι όσοι έχουν ανάγκη ε, μπορούν να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους σύρους αδελφούς μας και το 90% αυτό που βοηθούμε είναι μουσουλμάνοι και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Δεν το κάνουμε αυτό για διαφήμιση κάνουμε ό,τι μπορούμε, προσπαθούμε να ανοίξουμε ένα δρόμο για να μπορέσουμε ακριβώς να αντέξουμε. Σε όλα αυτά τα οποία είπα, σκοπός μου δεν ήταν ε, να φανούν σαν πολιτική πράξη, γιατί δεν είμαστε εμείς πολιτικοί. Τα είπα γιατί νομίζω ότι μας επιτρέπεται πλέον να πούμε ότι η οδύνη των σύρων πολιτών αξίζει να ενδιαφερθούμε για αυτήν. Αξίζει να ε, υπογραμμίσουμε αυτό τον ηρωισμό που επιδεικνύουν κάθε μέρα οι Σύριοι πολίτες, όλοι αυτοί τους οποίους βλέπει κανείς στους άδειους δρόμους της πόλης, που είναι σιωπηλοί, που έχουν εξαναγκαστεί στη σιωπή, που δεν μπορούν να εκφραστούν. Η πλειονότητα των Σύρων πολιτών δυστυχώ σιωπά σήμερα, δεν έχει φωνή για να αρθρώσει ε, τον πόνο της. Ο ηρωισμός τους λοιπόν αξίζει να υπογραμμιστεί όπως και η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη η οποία ξεπερνά τις διαχωριστικές γραμμές οι οποίες εκτείνονται και ξέρετε πολύ συχνά χωρίζουν ανθρώπους που η γεωγραφική τους απόσταση είναι μόνο ένα-δυο μέτρα, άντε τρία. Ε, δεν υπάρχει τίποτα πλέον να κάνει κανείς και γι' αυτό δεν αναζητώ να κάνω κάτι, δεν επιζητώ να κάνω κάτι, ούτε ελπίζω ότι θα λύσω το πρόβλημα. Όμως μαζί αυτό το οποίο ελπίζουμε είναι να μπορέσουμε να αντέξουμε για να βρούμε ένα νόημα, μια ουσία σε όλα αυτά, για να δείξουμε την αναγνώρισή μας έναντι όλων αυτών που μας εκφράζουν την αλληλεγγύη τους. Αυτό θα μας επιτρέψει να αντέξουμε και να αντισταθούμε σε αυτό το μεγάλο ε, πειρασμό του να αποθαρρυνθούμε και να μην βρούμε κανένα νόημα σε όλα αυτά και να τα παρατήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Χόφμαν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρευρεθώ σήμερα εδώ για να συζητήσουμε σε αυτό το πάνελ, αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Όπως ε, σας είπα, εργαζόμαι με το Middle East Concern, που είναι ένα δίκτυο που ιδρύθηκε πριν 24 χρόνια με στόχο να προωθήσει τη θρησκευτική ελευθερία και ελευθερία των τοπιθήσεων ε, στην περιοχή αυτή, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Οι κύριες δραστηριότητες μας έχουν να κάνουν ε, με τις χριστιανικές κοινότητες, αλλά φυσικά υποστηρίζουμε θρησκευτική ελευθερία και ελευθερία επιθήσεων για όλες τις θρησκευτικές κοινότητες ε, και πιστεύουμε ότι αν αντιμετωπίσουμε κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές κοινότητες θα βοηθήσουμε και τις υπόλοιπες κοινότητες που αντιμετωπίζουν παρομοιότητες παρόμοια προβλήματα. Αν δούμε την ε, περιοχή, οι χριστιανικές κοινότητες στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή ε, διαιρούμε συνήθως την περιοχή σε τρεις υποπεριοχές. Η πρώτη ε, θα ήταν ε, από τη Μαυριτανία ως την Τινσία, την Εμένη και την Αραβική Χερσόνησο και τη Σομαλία, ε, όπου εκεί έχουμε σχετικά μικρό αριθμό χριστιανών από κάποιες εκατοντάδες σε κάποιες χώρες μέχρι κάποιες δεκάδες χιλιάδες χώρες όπως η Αλγερία στο σύνολο της χριστιανικής κοινότητας θεωρείται ότι έχει αλεξοπιστήσει από το Ισλάμ ε, και το λέω αυτό γιατί κάποιοι τώρα είναι τρίτης γενιάς, δηλαδή οι παππούδες τους ε, είναι αυτοί που από το Ισλάμ άλλαξαν θρησκεία και πέρασαν στο χριστιανισμό και μεγαλώσαν τα παιδιά τους ως χριστιανούς. Τώρα είναι ενήλικα αυτά τα παιδιά και έχουν τα δικά τους παιδιά τα οποία τα μεγαλώνουν ως χριστιανούς, όμως όλες αυτές οι γενιές εξακολουθούν να θεωρούνται και από την κυβέρνηση και από την κοινωνία ότι έχουν εξοπιστήσει από το Ισλάμ. Η δεύτερη υποπεριοχή θα λεγόταν Κεντρική Μέση Ανατολή από το Σουδάν, την Αίγυπτο και κατόπιν προς το Βορρά καλύπτει όλες τις χώρες και την Τουρκία, Βόρεια και το Ιράν στα Ανατολικά. Οι χώρες αυτές έχουν μεγάλες ε, κοινότητες χριστιανικές, έχουν αναγνωριστεί από τις κυβερνήσει και υπάρχουν και κάποια δικαιώματα που τους έχουν δοθεί και υπάρχουν μικρό, υπάρχει μικρός αριθμός ατόμων που έχει στι χώρε αυτέ. αυτές και η τρίτη υποπεριοχή είναι η Αραβική Χερσόνησος, εκτός της Ιεμένης και η Λιβύη που έχουν μεγάλες θρησκευτικέ κοινότητε, αλλά κυρίως μιλάμε για εκπάτριδες. Πρόκειται για μετανάστες που δουλεύουν εκεί και υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα αναγνώρισης από τις κυβερνήσει στις χώρες φιλοξενίας. Τώρα, αν δούμε τα θέματα που οι χριστιανικές κοινότητες και άλλες μειονοτικές κοινότητες αντιμετωπίζουν, υπάρχει μια σειρά προβλημάτων. Δεν έχω φυσικά το χρόνο σήμερα το πρωί να αναφερθώ σε όλα εις βάθος. Απλώς ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε τρεις κυρίες κατηγορίες καταχρήσεων, παραβιάσεων των ανθρωπινών δικαιωμάτων και άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Το πρώτο, που μάλιστα είναι και στις ειδήσει αυτές τις μέρες, είναι η βία από τους μη κρατικού παράγοντες. Ήδη έχουμε ακούσει κάποια λόγια σχετικά από τον προηγούμενο μιλητή, ε, υπερισχύει σε διάφορες ε, καταστάσεις σειράξεων, στη Συρία φυσικά, Μόλις ακούσαμε ότι και στο Ιράκ έχουμε εξτρεμιστικέ ομάδε, όπως το Ισλαμικό κράτος, ε, ΔΕΣ ε, και άλλες διαπράττουν κτηνώδεις πράξεις ε, έναντι ανθρώπων οι οποίοι διαφωνούν μεταξύ τους φυσικά και κατά χριστιανικών κοινοτήτων και θα αναφερθούν και στο Ιράκ οι συνάδελφοι αργότερα. Αλλά αυτό το φαινόμενο δεν περιορίζεται απλά σε αυτές τις δύο χώρες. το χάρη, η Αίγυπτος έχει μακρά ιστορία βίας κατά των κοινοτήτων, κυρίως η Ανοαιγυπτός και σε μεγάλες πόλεις όπως την Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο έχουμε δει βία κατά ε, των χριστιανών, κατά των εκκλησιών, των ιδιοκτησιών τους και φυσικά και κατά ανθρώπων ορισμένες φορές. Συνήθως τα προβλήματα αυτά επιλύονται με το να ε, εξαναγκάζουν κάποιες επιτροπές συμφιλίωσης να συναντιούνται στα χωριά, στις κοινότητες και πολλές φορές κάποια άτομα θα πρέπει να δεκτούν ε, την ενοχή και πολλές φορές να πληρώσει κάποιο πρόστιμο ή κάποιος εκδιώκεται από το χωριό. Έχουν υπάρξει πολλές ε, τέτοιες περιπτώσεις στην Τουρκία και κυρίως ε, τα τελευταία χρόνια, μιλάμε για επιθέσεις κατά χριστιανών ή κατά ιδιοκτησία χριστιανών και πριν δύο μήνες ε, πυρπολήθηκε ένα κέντρο χριστιανών ε, στην Κωνσταντινούπολη και πολλά, πολλές από αυτές τις υποθέσεις ε, δεν ε, έχουν λυθεί, δεν έχουν αντιμετωπιστεί από τις αρχές επιβολής του νόμου και υπήρχαν και επιθέσεις και στη Λιβύη. Πριν μία εβδομάδα είχαμε και τον αποκεφαλισμό, αυτόν τον τρομακτικό αποκεφαλισμό 21 χριστιανών. Αυτό δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Πέρσι τουλάχιστον 24 ε, κόπτες της Αιγύπτου δολοφονήθηκαν στην Λιβύη αλλά και χριστιανοί από άλλες εθνικότητες ε, και δυτικοί επίσης δολοφονήθηκαν πέρσι στη Λιβύη. Και θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα. Στις περιοχές όπου υπάρχει αναγνωρισμένη εκκλησία από τις αρχές, εξακολουθούν να υπάρχουν ε, κάποια προβλήματα. Ένα πρόβλημα που συμβαίνει πολύ συχνά έχει να κάνει με τα κτίρια. Ε, με τις εκκλησίες ως κτίρια. Πολλές φορές υπάρχουν περιοριστικές κρατικές πρακτικές ε, ή νόμοι σε ό,τι αφορά το χτίσιμο των εκκλησιών και στην Αίγυπτο, παραδείγματο χάρη, χρειάζεται ειδική άδεια από τον πρόεδρο για να χτίσει κανεί μια νέα εκκλησία. Είναι πολύ δύσκολο να πάρει κάποιο αυτή την ε, άδεια και επίση ε, χρειάζεται και άδεια από άλλε αρχέ, κατώτερε αρχέ για επισκευέ. Και φυσικά η βία αυτή κατά το κυριοτήτων συνήθω ξεκινά από μια φήμη που διαδίδεται ότι οι χριστιανοί προσπαθούν να χτίσουν μια εκκλησία χωρί να υπάρχει άδεια από την κυβέρνηση. Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα παραδείγματα στο Σουδάν, λόγου χάρη. Η κυβέρνηση δημόσια έχει δηλώσει από το 2011 ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να χτιστούν νέες εκκλησίες. Συστηματικά ε, κλείνουν ε, τις εφιστάμενες εκκλησίες. Ε, το είδαμε αυτό στις 18 Φεβρουαρίου μάλιστα. Επίσης στην Τουρκία εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με την επιστροφή ή την έλλειψη της επιστροφής ιδιοκτησίας στην Εκκλησία και μάλιστα και κτηρίων που έχουν δημευτεί τα τελευταία χρόνια και είναι πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο να πάρει κάποιο άδεια για να χτίσει νέες εκκλησίες. Ένα άλλο προφανές παράδειγμα είναι στο Ιράν, όπου και πάλι η κυβέρνηση κλείνει όλα τα επίσημα εκκλησιαστικά κτίρια το τελευταίο έτος και μιλάμε για τρόπους ε, που συναντιούνται χρησιμοποιώντας τα φαρσί. Ενορίες που συναντιούνται μιλώντας τα φαρσί. Και επίσης στη Βόρεια Αφρική δεν ε, υπάρχει επίσημη αναγνώριση. Υπάρχουν μόνο λίγα κτίρια που έχουν αναγνωριστεί και έχουν καταγραφεί για τους ε, για τους μετανάστες, εκπάτριδες, ε, οι υπόλοιποι πρέπει να συναντιούνται κρυφά. Στην Αραβική Χερσόνησο έχουμε ε, συγκεκριμένα κτίρια και οι χριστιανικές κοινότητες συνήθως επιτρέπεται να αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους αν ε, δεν προβαίνουν σε πολιτικές ε, πράξεις ε, ή δεν επιτρέπουν σε μουσουλμάνους να έχουν πρόσβαση εκεί, αλλά το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πάρα πολύ λίγα τέτοια συγκροτήματα που έχουν σχεδιαστεί για να υποδεχτούν λίγες χιλιάδες ανθρώπους και ε, συνήθως πρέπει να χρησιμοποιούνται από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και επομένως υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν έχουν πρόσβαση και υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά όπου οι άνθρωποι απλώς επειδή δεν υπήρχε χώρος αποφάσισαν να υλοποιήσουν θρησκευτικές δραστηριότητε έξω από τα εκκλησιαστικά κτίρια και συχνά αντιμετώπισαν προβλήματα με τις αρχές επειδή είχαν θρησκευτικές συναντήσεις έξω από τα εκκλησιαστικά κτίρια. Και ένα τελευταίο παράδειγμα. Με αναφέρω και πριν σε όλες τις χώρες της περιοχής Έχουμε και χριστιανούς ε, από μουσουλμανικό παρελθόν ε, που οι παππούδες τους παραδείγματος χάρη είχαν ε, αποφασίσει να αλλάξουν θρησκεία και αντιμετωπίζουν μια σειρά προβλημάτων. Σε μεγάλο βαθμό δεν είναι αποδεκτή στην κοινωνία και συχνά τους απορρίπτει είτε η οικογένειά τους είτε η κοινωνία Μπορεί να πάρει αυτό πολλέ μορφέ, αλλά τουλάχιστον δεκάδε από αυτού ε, δολοφονούνται κάθε χρόνο. Δεν αναγνωρίζονται από τι κυβερνήσει. Και κάθε χρόνο έχουμε πολλέ περιπτώσει ανθρώπων ε, που συλλαμβάνονται. Πολύ λίγες ε, χώρες στην περιοχή έχουν την αποστασία ή το να αλλάξει κάποιος θρησκεία και να εγκαταλείψει το Ισλάμ ως έγκλημα πολλές φορές σε χώρες όπως το Ιράν, ε, όπου έχουμε ε, πάνω από 100 άτομα που έχουν ελαξοπιστήσει στη φυλακή και αυτοί έχουν καταδικαστεί ή κατηγορούνται για πολιτικά εγκλήματα ή για βλασφημία ή για άλλου είδους εγκλήματα που έχουν να κάνουν με τη θρησκευτική ελευθερία. Και ακόμη και αν δεν έχουν ε, διωχθεί ποινικά, εξακολουθούν ε, να υπάρχουν πάρα πολλές επιπτώσεις ε, σε προσωπικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά θέματα επιμέλειας, γάμου, κληρονομιάς, οικογενειακά ζητήματα δηλαδή όπου υπάρχουν ε, περιορισμοί για το ποιον μπορούν να παντρευτούν, αν έχουν παιδιά, πρέπει να μεγαλώσουν τα παιδιά τους ως μουσουλμάνους ε, και όταν ε, πεθάνουν πρέπει να θαυτούν σε μουσουλμανικά νεκροταφεία με μουσουλμανικές τελετές. Συχνά υπάρχουν ε, μέλη της οικογένειας, μουσουλμάνοι, που αρνούνται να τους οργανώσουν μία χριστιανική ή θρησκευτική τελετή. Και επίσης σε πολλές περιοχές, χώρες της περιοχής ε, διάφορες κοινότητες ε, έχουν ε, δική τους ενορία και έχουν δικά τους συγγνώμη δικαστήρια γιατί αν καταδικαστούν από τα κοινωνικά δικαστήρια ουσιαστικά πάβουν να υπάρχουν ως άνθρωποι με δικαιώματα. Αυτό αποκαλείται αστικός θάνατος δηλαδή οποιαδήποτε συμφωνία ή σύμβαση έχουν, έχουν συνάψει ακυρώνεται, δεν μπορούν να έχουν λογαριασμό στην τράπεζα, δεν μπορούν να έχουν ιδιοκτησία, ε, τους ε, αφαιρούν το διαβατήριο και φυσικά σταματούν να υπάρχουν ε, για οποιαδήποτε νομική συναλλαγή. Αυτό είναι λίγα παραδείγματα διαφόρων παραβιώσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ε, οι χριστίνικες κοινωνότητες και κατά επέκταση και άλλες ε, μειονοτικές κοινότητε στην περιοχή. Θα μπορούσα να έχω αναφέρει πολλά περισσότερα. Όμως νομίζω ότι αυτό που δείχνουν πολλά από τα παραδείγματα αυτά είναι ότι αν ε, και υπάρχει μεγάλη ένταση σήμερα απέναντι στις ε, τρομερές πράξεις που λαμβάνουν χώρα εντός του εμφυλίου ή από ομάδες όπως το Ισλαμικό κράτος και άλλους εξτρεμιστές ε, και φυσικά δίνεται πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτές τις κτηνοδίες. Όμως η παραβιαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων έναντι των χριστιανών ε, και άλλων κοινοτήτων δεν ξεκίνησαν με την έναρξη αυτών των σειράξεων ε, και την ανάδυση ομάδων όπως το Ισλαμικό κράτος. Αυτές οι παραβιάσεις δυστυχώς δεν θα σταματήσουν με το τέλος αυτής της σύνταξης ή με την ήττα του Ισλαμικού κράτους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να, Κύριε Χόφμαν και τώρα ο Βίλιαμ ε, διευθυντής του ε, Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους ε, όσοι βοηθήσατε στη διοργάνωση αυτής της ακρόασης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Υπόσχομαι να είμαι σύντομο. Ξέρω ότι έχετε επιδείξει πολύ μεγάλη υπομονή. Πολύ γρήγορα να σας δώσω ένα υπόβαθρο. ε, ε μεγάλη χαρά σας καλούμε να διαβάσετε τελευταία μας έκθεση. Στις συμπληγάδες ε, το, ε, η κατάσταση των μειονοτήτων στο Ιράκ μετά την πτώση της Μοσούλης. Έχουν γίνει διάφορα στρατιωτικές επιχειρήσεις και τα αλλά εμεί θέλουμε να σας δείξουμε τι έγινε στο Ιράκ για τις πιο ευάλωτες ευπαθείς ομάδες. Τέσσερις οργανώσεις με κυβερνητικές στο δικό μας Ινστιτούτο ε, έχουν συνεργαστεί για αυτή την έκθεση, το οποίο εγώ εκπροσωπώ, η ε, ε, Διεθνής Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων, η οργάνωση Όχι Ειρήνη Χωρίς Δικαιοσύνη και η οργάνωση των λαών και των εθνών που δεν εκπροσωπούνται. Υπάρχουν εδώ μερικές εκθέσεις στην είσοδο και σε κάθε ιστότοπο της κάθε μιας από τις οργανώσεις αυτές μπορείτε να βρείτε την έκθεσή μας. Σας παρακαλώ να τη λάβετε υπόψη. Γιατί το ονομάσαμε έτσι το έγγραφο αυτό ανάμεσα σε συμπληγάδες. Γιατί ακόμα και πριν ε, την ε, ε, ISIS στο Βόρειο Ιράκ το 2014 η κατάσταση των μειονοτήτων στο Ιράκ ήδη ήταν πάρα πολύ ικτρή, ιδιαίτερα εκεί που ζούσαν σε παιδινές περιοχές ανάμεσα σε δύο πυρά, Κούρδους και η Ιρακινή κυβέρνηση. Ακόμα και πριν πέσει η Μοσούλη περίπου οι μισή είχαν φύγει από τη χώρα από το 2003 και μετά. Και θέλαμε να πούμε ότι η κατάσταση ήταν κακή έτσι και αλλιώς που έχει χειροτερεύσει πάρα πολύ σήμερα. Και μετά το ISIS υπάρχει και μια νέα νοτροπία το Ισλαμικό κράτος. Χιλιάδες ε, ε, ήταν οι δολοφονίες, ακροτηριασμοί, απαγωγές, άγνωστος αριθμός γυναικών κοριτσιών που αναγκάστηκαν να παντρευτούν, έγιναν ε, σεξουαλικές κλάβες και δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ε, έχουμε καλύψει πάρα πολλά θέματα και η κατάσταση είναι πολύ ζωφερή. Ε, ακροτηριασμοί, ε, ε σεξουαλική βία, βασανιστήρια, συνοπτικές εκτελέξεις, ε, παιδιά, ε, είναι πράγματα φρικτά. Ας πούμε, ε, πολιτιστική και θρησκευτική ιδιοκτησία αιώνων έχει καταστραφεί και είναι ε, τρομερές οι ε, καταχρήσεις καθημερινά και φαίνεται ότι συνειδητά υπάρχει μια απόπειρα να εκριζωθεί η εθνική και θρησκευτική ε, πολυμορφία του Ιράκ. Μόλις εκτές διάβασα ότι στην Μοσούλη ε, γίνονται λαιλασίες και καίνε βιβλία από το ε, Πανεπιστημιακό ε, η Βιβλιοθήκη της Μοσούλης. Έχουν πάρει 8.000 βιβλία και τα καίνε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Θα πρέπει με την έκθεση αυτή να σας ενημερώσουμε και με κάποιες ιστορίες που ακούσαμε και είχαμε συνεντεύξεις με ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν. Ένα κορίτσι, Γεζιντή, 17 ετών, μας είπε, μια μέρα, τρεις η ώρα το απόγευμα, η οικογένειά μου πήγαιναμε σε ένα κοντινό χωριό και είδαμε μαχητές του ISIS που είχαν και σημαία ε, ε, Γεζιντή μας είπαν να μην κουνηθούμε και θα γυρίσουμε σπίτι μας αργότερα. Μετά από ε, λίγες ώρες, δέκα αυτοκίνητα ήρθανε και πήραν όλους τους άνδρες, τις οικογένειες και τους πήγαν στο βουνό και τους σκότωσαν. Πατέρα, αδέλφια, ξαδέλφια. Μετά ήρθαν και πήραν τους υπόλοιπους, τα κορίτσια. Ε, οχτώ παιδιά που ήταν μαζί μας, ε, ε ό,τι ε, όλους τους συγγενείς και μας πήγαν στην Ταλάφα όπου μείναμε για πέντε μέρες σε ένα σχολείο και δεν είχαμε καμιά επαφή με τους άντρες που μας απήγαγαν. Τους βλέπαμε μόνο όταν μας φέρνανε ε, τροφή και όταν βομβαρδίστηκε η περιοχή μας πήγαν σε άλλο σχολείο στη Μοσούλη που μείναμε άλλες πέντε μέρες. Μετά από άλλη αεροπορική επιτροπή μας πήγαν στη φυλακή της Μπατούς. Εκεί μας ε, ξεχώρεσαν από τα παιδιά που ήταν ηλικία 5 έως 10 ετών που τα πήγαν αλλού. Μείναμε δύο εβδομάδες και πλέον στη φυλακή και μετά μας ξαναπήγαν στο Ταλάφα όπου κορίτσια παντρεμένα και ανήπαντρα ε, ε, διαχωρίστηκαν. Μετά μας πήγανε στη Ράκα με την αδελφή μου σε ένα μεγάλο σπίτι με 100 άλλα κορίτσια. Ήταν ε, ένα παζάρι και 50 κορίτσια τα πούλησαν μέσα σε 5 μέρες και τις αδελφές μου που τις πούλησαν σε ένα Παλαιστινίο και ένα Ιρακινό στρατιώτη, μαχητή τους. Μας είπαν ότι θα μας πάνε στη Μοσούλη και η τιμή ήταν 1.000 ε, με 1.500 αμερικανικά δολάρια και τα ε, λεφτά ε, τα, τους έδινε ένας Σαβάραβας πρίγκιπας. Και είδα και στη Ράκα Ιρακινούς πώς καταλήγει αυτή η ιστορία. Αυτό το κορίτσι 17 ετών κατάφερε να ξεφύγει από τους ζημίους της και ξαναβρήκε την οικογένειά της και τώρα ε, μένει στην επαρχία Νταχούκ σε έναν καταβλισμό. Προσπαθώ να σκιαγραφίσω για να καταλάβουν οι πάντες ακριβώς τι συμβαίνει. Υπάρχει και μια άλλη όψη της που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Είναι όλες αυτές οι μετατοπίσεις, τα κύματα που έχουν προκύψει από τα εγκλήματα. Τα τελευταία ε, στοιχεία μιλούν για 2,5 εκατομμύρια ε, εκτοπισμένους σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Και βέβαια δεν έχουν τίποτα, ούτε έγγραφα, διαβατήρια, τους τα παίρνουν, ε, προσπαθούν να ξεφύγουν ε, από τις αιστείες τους και ζουν ε, διασπαρμένοι στην Ήπεθρο, κάτω από γέφυρες, σε γιαπιά, Υπάρχουν κάποιοι καταβλισμοί, αλλά είναι πραγματικά εκτρή η κατάσταση. Και η κατάσταση στους καταβλισμούς είναι πολύ χαμηλή, νερό δεν έχουν, δεν έχουν αποχέτευση, ε, ζουν σε σκηνές όταν υπάρχουν καταβλισμοί. Εμείς προσπαθήσαμε με την έκθεσή μας να τονίσουμε αυτό ε, και τα νομικά στοιχεία και τις πτυχές. Όταν μιλούμε για αυτή την κατάσταση, όλα αυτά τα εγκλήματα ε, του Ισλαμικού κράτους, ο κόσμος λέει είναι εγκλήματα πολέμου, είναι γενοκτονία και αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε και να συνεισφέρουμε προς την κατεύθυνση είναι να κάνουμε και μια νομική ανάλυση για όλες τις παραβιάσεις του ανθρωπίνου δικαίου ε, και τον, ε, ε, του διεθνούς δικαίου. Και σταματώ εδώ, θα δώσω το λόγο στην κυρία Άλισον Σμιθ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω. Όπως... Ε, είπε ο συνάδελφος για να εκπονήσουμε αυτή την έκθεση. Μελετήσαμε τι έγινε στο Βόρειο Ιράκ Ιούνιο με Αύγουστο του 2014 και τα είδαμε αυτά από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου, διεθνούς ποινικού δικαίου και ανθρωπιστικού δικαίου για να δούμε τι είδους εγκλήματα έχουν διαπραχθεί ενδεχομένω. Μπορείτε να δείτε στην έκθεσή μας ότι μπαίνουμε σε λεπτομέρειες για ειδικά στοιχεία για τα εγκλήματα και τις αξιόπινες πράξεις. Δεν θα μπω εγώ σε αυτό. Θα ήθελα να σας δώσω μια ε, συνολική θεώρηση ε, και το τι διαπιστώσαμε ως προς εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία. Εγκλήματα πολέμου, από τα γεγονότα που έχουμε από την έκθεση, έχουμε εντοπίσει ότι είναι μία διεθνής ένοπλη σύραξη στο Ιράκ τότε που σοβούσε και ακριβώς λόγω αυτού είναι 16 τουλάχιστον τα εγκλήματα πολέμου που ε, διεπράχθησαν τότε και μπορούμε να πούμε ότι οι ομάδες ε, ISIS ε, διέπραξαν 10 από τα 16 ας πούμε. Απαγή ομήρων, συνοπτικές εκτελέσεις, επίθεση σε κτίρια που ήταν κέντρα θρησκευτικά, ήταν νοσοκομεία ή πολιτιστικά κέντρα η ε, υποχρεωτική στρατολόγηση παιδιών κάτω των 15 ετών που συμμετέχουν ενεργά στις εχθροπραξίες. Από τις πληροφορίες που έχουμε μπορούμε να πούμε ότι φυσικά έχουν ε, διαπραχθεί εγκλήματα πολέμου. Σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ε, οι δυνάμεις του Ισλαμικού κράτους και συστηματικές και ευρείες επιθέσεις έχουν κάνει κατά των αμάχων στο Βόρειο Ιράκ. Το Διεθνές Δίκαιο επιβάλλει όταν υπάρχει τέτοια συστηματική, να μην υπάρχει συστηματική ή επανειλημμένη που υπήρξε ε, τέτοια επίθεση και έχουν διαπράξει 10 ε, από τις 11 απαγορευμένες πράξεις που συνιστούν ε, ε, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, δολοφονίες, σκλαβιά, βασανιστήρια, βιασμό, ε, δίωξη και απάνθρωπη ε, συμπεριφορά. Ο πλήρης κατάλογος είναι στην έκθεση. Βεβαίως έχουν λοιπόν διαπραχθεί και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όχι μόνο εγκλήματα πολέμου. Σε ό,τι αφορά τη γενοκτονία, βεβαίως σκοτώνουν, ακροτηριάζουν ανθρώπους και επιβάλλουν ε, συνθήκες διαβίωσης ε, για να εξορροθρευτούν ομάδες ολόκληρες. Βεβαίως ε, για να στοιχειοθετηθεί η γενοκτονία αυτό θα πρέπει να είναι εις βάρος προστατευμένων ομάδων με σκοπό να καταστραφούν και να εξαφανιστούν, να αφανιστούν ολοκληρωτικά. Βεβαίω έχει συμβεί αυτό και ε, σε προστατευμένε ομάδε εθνικέ και θρησκευτικέ μειονότητε στο Βόρειο Ιράκ και νομίζω ότι είναι σωστό να πούμε ότι αυτέ οι ενέργειε διαπράχθησαν και εσκεμμένω με ε, σκοπό ε, πλήρω ή εν μέρη να καταστραφούν αυτέ οι κοινότητε, να εξολοθρευτούν. Βλέπουμε ότι υπάρχει πρόθεση, φαίνεται αυτό από τη φύση των ενεργειών, από το είδο, από την κλίμακα, ας πούμε, προσιλητισμοί, εξαναγκαστικοί η ε, ε, τιμωρία ε, σε άμαχο πληθυσμό για, όταν μιλάει άλλη γλώσσα, τη δική του γλώσσα και τη δική του θρησκεία, το πολιτισμό ο πληθυσμός αυτός. Και προσπαθούν να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές κράτος, όπως ακούσαμε και προηγουμένως στη συζήτηση. Μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι υπάρχουν στοιχεία και στη γλώσσα των δικηγόρων που είμαι και εγώ ε, θα είναι υπόλογοι στη δικαιοσύνη για τα όσα πράττουν απέναντι στην ανθρωπότητα και ως προς τις γενοκτονίες στο βόρειο Ιράκ. Υπάρχουν ε, πολλά στοιχεία που το τεκμηριώνουν σε πολλές χώρες, σχεδόν σε όλο τον κόσμο και έχει σημασία να πούμε ότι μας κάνει εντύπωση στα εγκλήματα αυτά, όχι μόνο η κλίμακά τους, αλλά και η βιαιότητα, η ομότητα, ε, ο στιγνός χαρακτήρας, αλλά και ο συστηματικός ταυτόχρονα. Και είναι ε, όχι μόνο αδίστακτοι, αλλά καφιόνται κιόλα για τα όσα κάνουν. Ότι επιβάλλουν τον δρόμο ε, στο βόρειο Ιράκ, στον άμαχο πληθυσμό και σε άλλες χώρες, θριαμβολογούν και το επιδεικνύουν. Και δεν σας λέγω τίποτα καινούριο, δεν πρόκειται να σταματήσουν από μόνοι τους, εκτός αν τους σταματήσει κάποιος. Θα συνεχίσουν και θα συνεχίσουν να διαδίδουν πέρα από σύνορα, να, να αναπτύσσονται, προσπαθούν να επιβάλλουν ε, τρομοκρατία στο παγκόσμιο χωριό, ε, ε, με τον ίδιο τρόπο που τρομοκρατούν τα χωριά στο Βόρειο Ιράκ. Γι' αυτά τα πράγματα θα πρέπει να λογοδοτήσουν και θα πρέπει να αποζημιωθούν τα θύματα. Και ε, επειδή εγώ είμαι δικηγόρος και εσείς βουλευτές, οι κυβερνήσεις, μέλη της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να αναλάβουμε δράση για ειδικέ ε, συστάσεις θα, επανα... θα ξαναδώσω το λόγο στο ΣΠΕΝΣ. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που ξεπερνάω το χρόνο που μου έχετε δώσει, ωστόσο θα ήθελα να κλείσω με μια άλλη ιστορία ενός άνδρα γεζίδη 20 ετών που συναντήσαμε στους καταβλισμούς, τον ρωτήσαμε ποια είναι τα σχέδιά σου, τι θέλεις να κάνεις, ποιοι είναι οι στόχοι σου στη ζωή μακροπρόθεσμα και μας απάντησε. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα μας μεταφέρουν σε νέο καταβλισμό. Αυτό είναι το πρόβλημα με αυτή τη σκέψη οι εκτοπισμένοι δεν μπορούν να έχουν ορίζοντα, να έχουν μακροπρόθεσμη σκέψη και αυτό είναι σημαντικό. 38 βασικές συστάσεις έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επίκουσα ανθρωπιστική βοήθεια χρειάζεται. Το 36% ε, έχει δοθεί από το σύνολο ε, των ετοιμάτων για χρηματοδότηση από τα Ηνωμένα Έθνη μόνο και τα Ηνωμένα Έθνη και οι εκπρόσωποι τους μας απαντούν δώστε μας τα εργαλεία για να κάνουμε τη δουλειά και θα την κάνουμε. Αλλά ας μην υποκρινόμαστε ότι έχουμε τους πόρους ενώ δεν τους έχουμε. Έρευνα, διώξεις για τη διαφθορά στο σύστημα παράδοσης της ανθρωπιστικής βοήθειας. Όλα αυτά αναφέρονται στην έκθεση και το είπε και η Άλισον. Η δίωξη των εγκλημάτων που έχει διαπράξει το ISIS. Αναγνωρίζουμε ότι η μακροπρόθεσμη προεθεσμία και επανεγκατάσταση των εκτοπισμένων που ανήκουν στις μειονοτικές ομάδες θα πρέπει να εξεταστεί. Και αυτό που σας καλώ όλους να κάνετε είναι να αρχίσετε να κάνετε σχέδια για την εποχή μετά το ISIS. Το ISIS δεν θα είναι μεγάλη ανησυχία για πάρα πολλά χρόνια. Τελικά θα ε, νικηθούν. Ωστόσο πρέπει να έχουμε σχέδιο για το πώς θα καλυφθεί αυτό το κενό. Πρέπει να έχουμε ασφαλείς περιοχές για τις μειονότητες. Καμιά μειονοτική ομάδα δεν πρόκειται να επιστρέψει σπίτι της εάν δεν υπάρχει ασφάλεια στον τόπο αυτό. Αυτό είναι προϋπόθεση για οποιαδήποτε ρύθμιση ε, μακροχρόνια. Και πρέπει να δούμε και το θέμα της συμφιλίωσης, γιατί οι γείτονες αποφεύγουν γείτονες στη Μοσούλη. Πρέπει να γίνει συμφιλίωση σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο γειτονιάς. Και πρέπει να δούμε το θέμα της ανοικοδόμησης γιατί οι καταστροφές είναι τεράστιες. Όλα αυτά τα έχω αναφέρει στην έκθεσή μου. Θέλουμε να κάνουμε αυτή την παρουσίαση για να τονίσουμε το μέγεθος, των βεληνικές ε, ε, των προβλημάτων και των ε, ζητημάτων που μένει να ρυθμιστούν. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Και εγώ σας ευχαριστώ για να έχουμε μία άποψη του τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιες είναι οι κατευθυντηρίες γραμμές που ακολουθεί στον αγώνα για την θρησκευτική ελευθερία κατά των διακρίσεων και κατά ε, ε, της μυσαλλοδοξίας θα δώσω το λόγο στην κυρία Κάτεμπεργκ για λίγο από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί πρέπει να δώσουμε το λόγο και στους βουλευτές. Παρακαλώ κυρία Κάτεμπεργκ. Uh, ladies and gentlemen, για διακεκριμένα μέλη της ε, Επιτροπής αυτής θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Είμαι εκπρόσωπος του Open Doors International. Είναι μια οργάνωση που θέλει να βοηθήσει χριστιανούς όταν παραβιάζεται η ελευθερία πεπιθήσεων θρησκευτικών όχι μόνο των χριστιανών αλλά των πάντων. Και γι' αυτό είμαστε μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας ε, κατά της ε, θρησκευτικής μυσαλλοδοξίας και διακρίσεων. Και εκ μέρους αυτής της πλατφόρμας παίρνω το λόγο σήμερα. Θα ήθελα να σας κάνω μια σύντομη επισκόπηση του τι συμβαίνει. Η οργάνωσή μας ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό να βοηθήσει και να ανακοφίσει όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ε, θρησκευτικής και πίστης. Είναι η ΦΟΠ. Έχουμε ένα δίκτυο ε, διαφόρων οργανώσεων που είναι μέλη μας από ε, θρησκευτική ε, βάση αλλά και χωρίς θρησκευτική βάση. Θεωρούμε ότι η ελευθερία του θρησκεύματος συμβάλλει στη δημοκρατία, στην ανάπτυξη, στο κράτος δικαίου, στην ειρήνη, στη σταθερότητα. Είναι κάτι που διασφαλίζει την πολυμορφία. Έχουμε ε, τον ειδικό εισηγητή στη σχετική του έκθεση, τον κύριο Λαμπρινίδη, ο οποίος τότε στην έκθεσή του είχε υπογραμμίσει ότι ε, η ελευθερία του θρησκεύευστε είναι, ένα από τις, είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς λοιπόν δρούμε σε αυτό το πεδίο και ενθαρρυνόμαστε από τη διασφάλιση και την εγγύηση της ΥΠΑ της εκπροσώπου κυρίας Μογκερίνη, η οποία έχει υπογραμμίσει ότι η ελευθερία αυτή είναι αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής. Περιμένουμε τις στρατηγικές κατευθυντηρίες γραμμές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι είναι καλό το έγγραφο, πολύ εμπεριστατωμένο και, και μπορεί να ε, ξεδιπλώσει και να απομυθοποιήσει όλο αυτό το δικαίωμα της ελευθερίας του σκέπτεστε, του ε, θρησκεύεστε. Και μπορέσαμε εμείς να συμβάλλουμε σε αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης. Ε, στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ότι οι παραβιάσεις, οι καταστρατηγήσεις του δικαιώματος αυτού είναι πολύ ευρείες. Άκουσα τις ε, προηγούμενες παρουσιάσεις και συμφωνώ με τον κύριο Λαμπρινίδη απολύτως. Η πρόκληση μπροστά μας είναι πολύ σημαντική. Όμως οι κατευθυντήριες γραμμές είναι πολύ καλή βάση και δεν θα πρέπει να περιοριστούν μόνο επί χάρτου, θα πρέπει να μεταφραστούν στην πράξη, στην πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της. Οι αξιωματούχοι που είναι, λειτουργούν και δουλεύουν στις πρωτεύουσες αλλά και επί τόπου πρέπει να καταλάβουν τη δυναμική της ελευθερίας του θρησκεύεστε μέσα στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ποια θέση πρέπει αυτό να καταλάβει στο παγκόσμιο πολιτικό γίγνεσθε γιατί τελικά αυτοί θα το εφαρμόσουν επί τόπου. Χαιρόμαστε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, περιλάβει κατάρτιση για το δικαίωμα αυτό, την ενθαρρύνουμε να το συνεχίσει, να έχει ακόμα μεγαλύτερη κατάρτιση και εκπαίδευση να την προσφέρει στο προσωπικό της και ξέρετε, η κατάρτιση δεν είναι αυτός σκοπός, είναι ο καρπός, το αποτέλεσμα της κατάρτισης που θα διασφαλίσει την επιτυχημένη υλοποίηση των κατευθυντηρίων γραμμών. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι οι κατευθυντηρίες γραμμές είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα, δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Και θα ήθελα να σας δώσω κάποιες συστάσεις που συνάδουν με τις κατευθυντηρίες γραμμές με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή είναι ευθύνη των κρατών να διασφαλίσουν ότι τα άτομα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους να πιστεύουν ε, ελεύθερα σε όποιο δόγμα θέλουν, σε όποια θρησκεία θέλουν. Είναι πολύ σημαντικό η διεθνής κοινότητα, η ΕΕ, οι αρχές, τα σχετικά μέρη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή να καταδικάζουν και να συνεχίσουν να καταδικάζουν τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων αυτών ε, και θα πρέπει οι πολίτες να καθησυχάζονται ότι όσοι καταστρατηγούν τέτοια δικαιώματα δεν θα χαίρουν ατιμορρησίας. Ξέρετε, η κοινωνία της Μέσης Ανατολής απαρτίζεται, είναι ένα μοσαϊκό εθνοτικών κοινοτήτων και θρησκευτικών κοινοτήτων. Ωστόσο, μέρος της Μέσης Ανατολής ε, είναι στο χείλος της απώλειας της ποικιλομορφίας της. Μέχρι τα τέλη του 2014 το 40% των χριστιανών της Συρίας είχαν εγκαταλείψει τη χώρα. Αλλά και στο Ιράκ ε, υποδουλώνονται ή σκοτώνονται μέλη των μειονοτικών ομάδων και κοινοτήτων στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τη χώρα. Και ε, βλέπετε ότι είναι πολύ ανησυχητικό το τι θα συμβεί μέσα σε 20 χρόνια και μετά από 20 χρόνια. Είναι σημαντικό και στη Συρία και στο Ιράκ και στη Μέση Ανατολή να τονίσουμε ε, την αξία, τη σημασία αυτών των αξιών και να προωθήσουμε την ποικιλομορφία, την ισότητα για όλους. Και θα ήθελα να τονίσω ότι η εξωτερική πολιτική της ΕΕ, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία του θρησκεύεστε δεν θα πρέπει να έρχονται να επικαθίσουν ε, πάνω σε ένα καθεστώς σχετικής σταθερότητας άπαξ και αυτό επιτευχθεί. Αντίθετα, οι στρατηγικές που στοχεύουν στην πρόληψη των συγκρούσεων, στη διαμεσολάβηση, στην οικοδόμηση της ειρήνης πρέπει εγγενώς να περιλαμβάνουν αυτή τη διάσταση, αυτό το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας. Ξέρετε, πολλοί ηγέτες Άραβες έχουν, ε, τα, έχουν ταχθεί υπέρ της ποικιλομορφίας αυτής, της ε, δυνατότητας και σε τοπικό επίπεδο γίνονται προσπάθειες για συμφιλίωση στην Μέση Ανατολή. Ενθαρρύνω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, είναι πολύ συγκεκριμένες και έχουν αναλυφθεί πρόσφατα, να ενθαρρύνει τη συζήτηση, το διάλογο για το ρόλο που μπορούν να ε, διαδραματίσουν οι θρησκευτικέ κοινότητες και οι οργανώσεις που βασίζονται στη πίστη, στο δόγμα. Πώς μπορούν να συμβάλλουν δηλαδή στη συμφιλίωση, στην οικοδόμηση της ειρήνης. Ε, η οργάνωσή μας, η ΦΟΠ, έχει να κάνει, προβάλλει το δικαίωμα για όλους, για όλους τους ανθρώπους. Είναι θεμελιώδες στη δημοκρατία, είναι θεμελιώδες στον πλουραλισμό και στη διατήρηση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, να μπορεί κανείς να έχει ελευθερία του θρησκεύεστε. Σε όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η σημασία τους μπορεί να τονιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τη δική σας υποεπιτροπή. Ε, χαιρόμαστε διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δημιουργήσει την ομάδα για την ελευθερία του θρησκεύεστε και την ανεξιθρησκεία, την ενδιάμεση ομάδα ε, Intergroup, κομματική και ε, δεν θα πρέπει βέβαια μόνο η ομάδα αυτή να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Ε, νο, τα μέλη, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ασχοληθούν με αυτό το θέμα, να διερευνήσουν τις παραβιάσεις ε, με συζητήσεις, με εκθέσεις αναχώρα, με αντιπροσωπείες, με αποστολές, με ψηφίσματα και ε, θεωρούμε σε κάθε περίπτωση ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση αυτών που αλλαξοπιστούν. Όσοι τελικά ε, αλλάζουν δόγμα, υφίστανται πάρα πολλές συνέπειες και καλούμε την Επιτροπή σας να παρακολουθεί στενά τα, ε, την κατάσταση αυτή, αυτών των ατόμων και την εξέλιξη της νομοθεσίας για τη βλασφημία και για την αποστασία. Θέλουμε να εκφράσουμε τη στήριξή μας στο πρόσφατο κάλεσμα της διακομματικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ελευθερία του θρησκεύεστε κατόπιν ε, ε, σύστασης της κυρίας Αμογκερίνη της ΥΠΑ εκπροσώπου. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερο και συμφωνούμε με αυτό για να καταπολεμηθούν οι διώξει ανθρώπων που είναι άθεοι ή που έχουν μια ουμανιστική ε, αντίληψη του κόσμου και πεποίθηση του κόσμου. Και τέλος, ως προς τα δικαιώματα των γυναικών, ενθαρρύνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενσωματώσει και αυτή τη διάσταση της θρησκευτικής ε, ελευθερίας και άνεξη θρησκείας κάθε φορά που συζητείται το θέμα των ε, δικαιωμάτων των ε, γυναικών. Άλλωστε, το θρήσκευμα των γυναικών ενδεχομένως είναι το εκάστοτε είναι που τις κάνει ακόμα πιο ευάλωτες σε περίπτωση συγκρούσεων, ενόπλων συγκρούσεων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά γιατί προσκαλέσατε την οργάνωσή μας σήμερα εδώ. Έχουμε περιγνωμοσύνη για όλα αυτά τα θέματα και με χαρά θα τα συζητήσουμε κάθε φορά με εσάς. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ να δώσω την Προεδρία ε, στην ε, κυρία Μαρίσα Ματίας, η οποία ε, θα προεδρεύσει στο τέλος της συνεδρίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα περιμένω να βάλετε και ακουστικά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους και όλες ε, που μας ε, αφηγήθηκαν τόσο σημαντικά σε αυτή τη συνεδρίαση. Έχουμε αυτή την κοινή συνεδρίαση τώρα μεταξύ της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της ε, Αποστολής για τις χώρες του Μασρέκ. Φυσικά δίνουμε πολύ μεγάλη προσοχή και στην Επιτροπή και στην Αντιπροσωπεία και φυσικά θέλουμε να μην έχουμε κατακαιρματισμένη συζήτηση, θέλουμε να ενώσουμε τις προσπαθίες μας και να προσπαθήσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ενισχυμένες και ενοποιημένες συζητήσεις σε αυτόν τον οίκο. Εμείς είχαμε προγραμματίσει αυτή η συνεδρία στην διαρκέση μέχρι τις 11.30 και βέβαια τώρα όμως ε, υπάρχει μια γενοδορία από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μπορούμε να πάμε μέχρι τις 12. Όμως θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδελφούς να είναι όσο δυνατόν πιο σύντομοι ε, στις παρεμβάσεις τους και αν έχουμε δυνατότητα θα ακούσουμε και τους εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ τώρα έχω δύο συναδέλφους εδώ γεγραμμένους που έχουν ζητήσει το λόγο και Νομίζω ότι όταν θα μιλάω πρώτα συνάδελφο, θα ζητήσουν και οι υπόλοιποι που επιθυμούν το λόγο. Καταρχήν ο κύριος Βάιντασον. Ο κύριος Βάιντενχόλτσα. Ε, δεν είχα καταλάβει. Βάιντεν Χόλτσερ λέγομαι. Εντάξει. Ε, δεν κατάλαβα πολύ καλά το όνομά μου. Ε, Τρία πράγματα, πολύ σύντομα. Τώρα τι γίνεται. Αυτό τον καιρό. Στο Βόρειο Ιράκ ακούσαμε ότι έχουν συλλάβει, έχουν απαγάγει 200 ασύρο χαλδαίους τώρα στο Βόρειο Ιράκ. Και τι γίνεται με αυτούς. Η συνάδελφος Άννα Γκόμες και εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι ε, μετέβημεν στο Βόρειο Ιράκ. Συζητήσαμε και με γεζιτή οι ίδιοι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που είναι στα νύχια του Ντάεσ. 3.000-4.000 γυναίκες ε, είναι ιδιοκτησία, το λέω συνειδητά, ιδιοκτησία τους, κτήμα τους έχουν αγοράσει. Συζητάμε ολόκληρη την περιοχή, αλλά ερωτώ, γιατί δεν μπορούμε να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση σε χώρες με τις οποίες έχουμε κανονικές σχέσεις και έχουμε συζητήσει με γυναίκες και γνωρίζουμε γιατί μας είπαν ότι οι αδερφές τους, οι γειτόνισσες είναι ήδη στη Σαουδική Αραβία. Γιατί τις αγόρασε ένα Σαουδάραβας και είναι στο έλεος τους. Για τους καταβολισμούς των προσφύγων, το είπατε και εσείς, είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχουν χρήματα γενικά. Ε, οι πόροι που αφιερώνουμε εκεί είναι γελοί ε, λόγω τη καταστροφή και δεδομένη τη κατάσταση, Έχω πάει και εγώ σε προσφυγικό καταβλισμό. Ξέρετε, όταν πηγαίνει μια αντιπροσωπεία γίνεται μεγάλη φασαρία, έρχεται κόσμο, έρχεται ένα νέο και μιλάει αγγλικά και του λέω γιατί μιλά αγγλικά. Λέει βρήκα ένα λεξικό και μαθαίνω αγγλικά από το λεξικό. Ε, αν αυτό είναι ο μόνο τρόπο να κάνουν μάθημα στου καταβλισμούς, να πηγαίνουν σχολείο, τι θα γίνουν σε δύο, τρει, τέσσερι πέντε μήνε. Έχουν τόσο χρόνο εκεί ελεύθερο, δεν ξέρουν τι να τον κάνουν. Τι θα απογίνουν αυτά τα παιδιά. Έχουμε ανάγκη μεγάλη από πολλά περισσότερα χρήματα. Νομίζω συνολικά 60 εκατομμύρια ευρώ είχαμε. Μα πραγματικά είναι γελία τα λεφτά αυτά ε, και θαυμάζω τους ε, επαγγελματίε που εργάζονται εκεί, αλλά δεν φτάνουν ούτε για ζήτο αυτά τα λεφτά. Γιατί είναι πάνω από εκατομμύριο αυτοί οι άνθρωποι. Ε, και για την κατάσταση μετά το, το ISIS, ε, χαίρομαι που το αναφέρετε έτσι γιατί χρειάζεται και αισιοδοξία για να φτάσει κανείς ε, να σκεφτεί την κατάσταση μετά. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι σημαντικό και θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Ε, επανειλημμένα ακούστηκε η συμφιλίωση και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Κάτι που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση οι άνθρωποι αυτοί ζουν στην περιοχή από την εποχή του Χριστού. Τι θέλουμε, να φύγουν όλοι οι χριστιανοί από εκεί και να πούμε ότι ελάτε όλοι σε εμά. Ή μήπως θα πρέπει να ενδιαφερόμαστε να παραμείνει και ο χριστιανισμός που είναι τμήμα αυτού του ψηφιδωτού και τη πολυπολιτισμική κοινωνίας της Ανατολής. Ε, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, θα εξαφανιστούν οι χριστιανοί. Ευχαριστώ. Γιάννα. Κυρία Γκόμες όπως είπε και ο Τζότζεφ, τους περασμένους μήνες ε, εμείς ε, ταξιδέψαμε του Αγγλιστοκυρκού και συζητήσαμε με θύματα των μηνοτήτων ήταν πραγματικά συγκινητικό όχι μόνο ακούσαμε πολλά από τα θύματα, πολλές μαρτυρίες, όπως αυτές που διάβασε ο κύριος Σπένσερ και όλοι φυσικά έκλαιγαν στην αίθουσα. αλλά μιλήσαμε και με άλλους εκπροσώπους ε, των κοινοτήτων, ε, επισκεφτήκαμε καταβλισμούς και οργανωσμένους αλλά και άτυπους ε, και το συμπέρασμά μου είναι... Μάλλον γράψαμε και μια επιστολή στην κυρία Μογκερίνη και το συμπέρασμα είναι ότι δεν επαρκεί το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αρρωγή που προσφέρει στα θύματα και φυσικά τώρα έχει επιδεινωθεί η κατάσταση από το Ισλαμικό κράτο, αλλά ήδη ήταν πολύ άσχημη η κατάσταση με του Γεζίτη. Επισκεφτήκαμε την κοινότητα αυτή και μας είπαν ότι ήταν θύματα μιας ε, σφαγής ε, από την επίθεση στα βουνά τους ε, το περασμένο καλοκαίρι. Είναι η 22η σφαγή στην ιστορία. Η 72η σφαγή στην ιστορία, 22 η ένα ζωτικό θέμα ήταν το εξής. Πέρα από τα χρήματα είναι το να βοηθήσουμε τις ομάδες για να συνδράμουν ε, στο να σωθούν τα κορίτσια που κρατούνται όμοιροι. Εμείς μιλήσαμε με κορίτσια που μπόρεσαν να το σκάσουν, ε, γιατί υπήρχε ένα δίκτυο ε, και μάλιστα και κάποιες από τις γυναίκες που δούλευαν με το Ισλαμικό κράτος τους βοήθησαν να ξεφύγουν, είναι δυνατόν. Αυτή θα πρέπει να είναι μία από τις προτεραιότητές μας, να συστήσουμε εκεί τοπικές ομάδες με εντόπιους για να μπορούν να πάνε να βοηθήσουν και να σώσουν τις γυναίκες και τα παιδιά. Μιλήσαμε με πολλές γυναίκες, μας έδειξαν τις φωτογραφίες των νερών αδελφών τους. Ε, και ε, ξέρετε ότι στα στα μέσα κοινωνική δικτύωσης γίνεται πλήση εγκεφάλου εκεί από τους ισλαμιστέ. Και φυσικά υπάρχει και το θέμα της πολιτικής και δεν θα μιλήσω τώρα εδώ για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συντονίζει τα κράτη-μέλη, γιατί τα κράτη-μέλη δεν επιτρέπουν ε, σε αυτού τους να συντονιστούν ε, σε ό,τι αφορά το χάρη τη στρατιωτική στήριξη στους Πεσμεργά που πολεμούν του τρομοκράτε. Δεν μιλώ για την ε, ανθρωπιστική συνεργασία που θα έπρεπε να υπάρχει μεταξύ την, ε, της ε, ΕΚΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ικανοί άνθρωποι στο Ερμπίλ, αλλά δεν ξέρουν τι ακριβώς κάνουν τα κράτη-μέλη, ακριβώς στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, στον ίδιο τομέα. Και για την βοήθεια, όπως είπε ο Τζότζεφ, δεν υπάρχουν σχολεία στους καταβλισμούς. Χιλιάδες παιδιά, αλλά δεν υπάρχουν σχολεία, είτε μιλάμε για χριστιανικού καταβλισμού, είτε για καταβλισμού με γεζίδι. Δεν υπάρχουν σχολεία. Και πριν μια εβδομάδα ήμουν στο Λίβανο και προσπαθήσαμε εκεί να συζητήσουμε το θέμα τη κρίση στο Λίβανο και στην Ιορδανία. 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες είναι στο Λίβανο, 385.000 παιδιά σε σχολική ηλικία και από τα οποία 400.000 δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Αυτό σημαίνει πως όχι μόνο δεν θα είναι ποτέ σε θέση να συμβάλλουν στην ενοικοδόμηση της χώρας τους ε, να επιστρέψουν, αλλά είναι ε, και ευάλωτα απέναντι στους τρομοκράτες. Δηλαδή δεν μιλάμε μόνο απλώς για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά μιλάμε για θέματα ασφάλειας, να έχουμε μια προοπτική τη ανθρώπινη ασφάλεια και τη δική μα ασφάλεια για να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Το σχολείο είναι κάτι πολύ ζωτικό και είναι μεγάλη αποτυχία του ΟΗΕ, δική μα επίση. Επίση, πολιτική θεωρήσεων. Χριστιανοί στο Ιράκ, ιερεί, ε, αρχέ αρχές στη χώρα, στο Ιράκ, μα είπαν μην ε, δημιουργείτε αυτά τα ηλίθια προγράμματα θεωρήσεων για χριστιανούς όπως κάνουν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί αυτό επιδεινώνει την κατάσταση. Δεν προσπαθούν απλώς ε, να σώσουν του ανθρώπου, αλλά να σώσουν του προσλαμιστικού πολιτισμού. Και αν κάποια κράτη-μέλη συστήνουν προγράμματα για του χριστιανού, ενώ θα έπρεπε να συστήσουν προγράμματα για τι γυναίκε, παραδείγματο χάρη, που χρήζουν ειδική ε, θεραπεία, αυτέ που έχουν δραπετεύσει από τη σκλαβιά. Σε αυτούς τους ανθρώπους ε, πρέπει να δίνονται θεωρήσει και θεραπεία όχι μόνο στους χριστιανούς, γιατί αυτό φυσικά θα, αυτό θα ενθαρρύνει τη χριστιανική κοινότητα που πιστεύει ότι δεν έχει μέλλον στο Ιράκ αυτή τη στιγμή να έρθει και θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Αν πράγματι δεν υπάρχει προοπτική να μείνουν εκεί, θα έρθουν στην Ευρώπη. Αυτή η προοπτική για το μέλλον στο Ιράκ απαιτεί όχι μόνο ε, να ιδρυθούν σχολεία και άλλες τέτοιες πολιτικές, αλλά να έχουμε και ένα μακροπρόθεσμο όραμα ασφαλές ε, μέρος να γίνει το Ιράκ. Επίσης, ε, αν δεν υπάρχει ασφάλεια, κανείς δεν θα επιστρέψει στην πόλη του αν δεν υπάρχει δίθυμης προστασία. Τώρα το να περιμένουμε ότι τα πράγματα θα επιδεινωθούν όταν θα υπάρχει πτώση της Μοσούλης, γιατί υπάρχουν και μεγάλα αισθήματα μνησικασίας ε, έναντι ε, των Σουνιτών που από την Χάνη να είναι και μειοψηφία στο Ιράκ και φυσικά γι' αυτό υποστήριξαν ε, το ISIS, αλλά έχουν μείνει με το ISIS ε, στη Μοσούλη και όταν θα αποσυρθεί το Ισλαμικό κράτος από τη Μοσούλη, τότε θα υπάρχουν αντίπεινα κατά των Σουνιτών. Έτσι λοιπόν η ανθρωπιστική κρίση θα επιδεινωθεί. Και Φυσικά οι άνθρωποι δεν θα επιστρέψουν ε, όπου ήταν πριν αν δεν έχουν διεθνή προστασία. Και ε, αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στην πραγματική προσπάθεια για συμφιλίωση. Πρέπει να υπάρχει πραγματική προσπάθεια συμφιλίωση. Επίσης, για ε, ε, τις κουρδικές αρχές, ε, οι κουρδικές αρχές υλοποιούν μια εκστρατεία για να ε, υπάρχει ε, δίκη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο του Ισλαμικού κράτους ε, και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το υποστηρίξουν αυτό και οι Ιρακινές αρχές. Είναι σημαντικό για όλες τις μειονότητες στο Ιράκ και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερη δουλειά σε όλες αυτούς τους τομείς και σε πολλούς άλλους που δεν έχω χρόνο να αναφέρω. Ευχαριστώ κύριο Στάνοκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, προς πρόσφατος αποκεφαλισμός των 21 κοπτών χριστιανών στη Λιβύη και ε, η απαγωγή των ε, Ασσύριων ε, στη Σύρια είναι άλλα κεφάλαια μια τραγωδία που εκτελήσεται στη Μέση Ανατολή και στη Βορειοαφρική Αφρική, κυρίω μετά από την εισβολή του Ισλαμικού κράτου στο Ιράκ. Υπάρχει συστηματική στρατηγική από τι τζιχαντιστικέ Ισλαμιστικέ ομάδε να απελευθερώσουν την περιοχή αυτή από τι μειονότητε, ιδίως από τους χριστιανούς. Όμως πρέπει να θυμόμαστε ότι φέτος είναι η εκατοστή επέτειος της γενοκτονίας των Αρμενίων. Όταν είχαμε συστηματική προσπάθεια από την ε, Οθωμανική Τουρκία ε, να σφαγιάσει και τι χριστιανικές μενότητε Σφαγιάστηκαν και Έλληνες αλλά και Ασσύριοι. Πάρα πολλοί σφαγιάστηκαν το 1915 και πόντι. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι έχουμε πογκρόμ κατά των χριστιανών ε, και άλλων μειονοτήτων στην περιοχή, αλλά το Ισλαμικό κράτος ε, αποτελεί ένα συνδυασμό της τρομακτικής ε, δίωξη ε, που λάμβανε χώρα κατά των εναρτηρίων πριν μία δεκαετία, κυρίως από την Αλκάιντα. Αλλά μιλώντας ως πολιτικός, ε, εγώ έθεσα τα δεινά των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη Μέση Ανατολή και το Πακιστάν από τότε που πρωτοεξελέγει εδώ πριν από μία δεκαετία. Όμως, ακόμη και η ομάδα στην οποία ανήκα τότε, το ΕΛΚ, που ονομάζεται για Χριστιανοδημοκράτες, ε, και ε, τότε, αν και παρουσιάζονται σε βεστή, δεν ήθελαν καν να κυρώσουν το έτοιμά μου να συζητήσει το θέμα. Έτσι λοιπόν χαίρομαι που τώρα όλες οι ομάδες, ακόμη και ομάδες από την αριστερά, ε, που ε, ε, καταλήγουν τώρα να θεωρούν ότι αυτό το θέμα είναι ζωτική ε, σημασία. Επίση, θυμάμαι ότι ο Επίτροπο πριν 10 χρόνια ζήτησε χρήματα για να βοηθήσουμε του Συρίου και την κυρία Γιαμπάσκοβα, την πρέσβυρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ιράκ. Όμω δεν υπήρχε απάντηση και έπρεπε να βασιστούμε σε ιδιώτε δωρητέ ολοκληρωτικά. Και όπω είπε και η κυρία Γκόμε, η κυβέρνηση Αλ Μαλίκη έχει ενδιαφέρον να προστατεύσει τους χριστιανούς στο Ιράκ και καθώς ε, ήμουν και πρόεδρος ε, της ομάδας φιλίας με το Κουρδιστάν, το κοσμική κυβέρνηση του Βορείου Ιράκ ήταν πολύ πιο γενναιόδορη στο να προστατεύσει ε, τους εσωτερικά εκτοπισμένους κυρίως ε, τους Γεζίντι και τους ε, χριστιανούς. Όμως ε, νομίζω ότι και η μόνη λύση είναι να σταματήσουμε το Ισλαμικό κράτος ξαφνικά. Δεν θα μεταμορφωθούν σε καλούς. Έχουμε τον υφιστάμενη συμμαχία, όμως μόνα τα εναέρια χτυπήματα, τα εναέρια πλήγματα δεν θα αρκέσουν. Θα πρέπει να ε, υπάρχει και συμμετοχή των περιφερειακών δυνάμεων, αλλά θα πρέπει να ασκήσουμε και πίεση στο Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία και ιδίω στο Κατάρ, στα κράτη του κόλπου. Το Κατάρ ε, είναι μεγάλο επενδυτή στην περιοχή και ευχαρίστω ε, θέλουν να επιτρέπουν τη χρηματοδότηση εκτρεμιστικών ομάδων στη Συρία και φυσικά και η Τουρκία, η οποία έχει στρίψει αλλού το πρόσωπό της και κάνει ότι δεν βλέπει τι συμβαίνει στη στη Συρία. Εν τω μεταξύ, φοβάμαι που λέω ότι, λυπάμαι που λέω ότι πραγματικά σφαγιάζονται συχνό γυναίκες και παιδιά από αυτούς τους φανατικούς. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε. Θα ήθελα να κάνω ένα γενικό σχόλιο σε σχέση με τα όσα μόλις είπατε για το ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον πολιτικών ομάδων. Ε, συγγνώμη που το κάνω εγώ. Είναι προσωπικό αυτό. Τώρα λέτε ότι μέχρι και αριστερά έχει ξυπνήσει και ενδιαφέρεται. Πρέπει να σας πω ότι ανέκαθεν ενδιαφερόταν η αριστερά για αυτό το θέμα. Μπορεί να έχουμε διαφορετικό τρόπο να το προβάλλουμε ή να το πλαισιώνουμε ε, αυτό το ενδιαφέρον. Δεν σημαίνει ότι αδιαφορούμε ε, για όλες τις ευάλωτες ομάδες ε, ενδιαφερόμαστε. Είτε είναι πολιτικό το θέμα είτε θρησκευτικό Πάντα εμείς το βλέπουμε έτσι και δεν ε, αγνοούμε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διάφορες ε, θρησκευτικές μειονότητες κτλ. Υπάρχουν και πολιτικές διαστάσεις όμως, δεν είναι μόνο οι θρησκευτικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές που αφορούν και τους άλλους κατοίκους των χωρών αυτών. Δεν μπορούμε να θεωρούμε τη θρησκεία ως το βασικό στοιχείο της ταυτότητας κάποιου. We ε, ε, ε, λοιπόν για όλες τις μειονότητες και τις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. Νέκαθεν ναι, ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Το θέμα είναι σε ποιο πλαίσιο το βάζεις. Ωραία. Ο κύριος Γκζίπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης, στη συζήτηση. Είναι πάρα πολύ σημαντική για μένα εγώ το είχα ζητήσει και χάρηκα πάρα πολύ που οι συντονιστές και όλες οι πολιτικές ομάδες με υποστήριξαν σε αυτό μου το αίτημα. Θα ήθελα να το υπογραμμίσω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, χαίρομαι ιδιαίτερος που εκπροσωπείται εδώ και η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις χώρες μας ΡΕΚ. Είναι πάρα πολύ σημαντική η αντιπροσωπεία για όλα τα θέματα που μας απασχολούν αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τους προσκεκλημένους ομιλητές μας, ιδιαίτερα τον ε, πατέρα Ναβράς Σαμούρ. Σας ευχαριστώ πολύ διότι εσείς ζείτε από πρώτο χέρι καθημερινά επί τόπου όλες αυτές τις θηριωδίες. Στα τέλη του 2008 ήμουν στη Συρία. Όχι μόνο στη Δαμασκό, επισκέφτηκα και άλλες περιοχές, ιδιαίτερα ε, παραμεθόριες και είχα την ευκαιρία να δω και εγώ από πρώτο χέρι την κατάσταση που επικρατεί εκεί προσφυγικούς καταβλισμούς. Τότε ήταν Παλαιστίνη από την προηγούμενη σύραξη. Επίσης συναντήθηκα και με εκπροσώπους της χριστιανικής μειονότητας στην Συρία κατόπιν ε, δικού μου αιτήματο. Ήθελα να τους συναντήσω, να τους ρωτήσω για το πώς ε, συμβιούν εκεί και ε, ποια είναι η συνύπαρξη με τις άλλες κοινότητες. Και πρέπει να σας πω ότι η εικόνα που μου έδωσαν τότε ήταν θαυμάσια, αν τη συγκρίνουμε με τη σημερινή βέβαια, αλλά ακόμα και τότε ένας από τους εκπροσώπους της, κάποιας χριστιανικής εκκλησίας μου είπε Ναι. Αυτό πια είναι παρελθόν, γιατί άλλαξε η κατάσταση έκτοτε. Και ε, τώρα έχουμε περιέλθει στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Όταν είχαμε αυτή τη συζήτηση το 2008, ουδής θα μπορούσε να φανταστεί και να προβλέψει πόσο ικτρή θα ήταν σήμερα η κατάσταση και ε, από πλευρά ανθρωπιστικής κρίσης. Οι μισοί περίπου έχουν πεθάνει ή είναι αγνοούμενοι ή έχουν μεταναστεύσει ή δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Ξέρουμε που βρίσκονται εσωτερικά εκτοπισμένοι. Ωραία, αλλά βλέπει και πόσοι είναι για να καταλάβει κανείς τι διάσταση έχει όλη αυτή η τραγωδία και το τράμα. Υπάρχει και κάτι ακόμα που νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο τελικά να ξεπεραστεί. Προφανώς ελπίζουμε οι σημερινοί δράστες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και αν κερδίσουμε θα επανέλθει η νομιμότητα. Ποια είναι η νομιμότητα και πώς επανέρχεται. Σας το δείχνει αυτό η ίδια η Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Πόσο δύσκολο είναι να ανοικοδομήσει κανείς τη χώρα του. είναι μια ενοπλή σύραξη αυτή που σοβεί εκεί με διαφορετική ε, κατάσταση και ως προς την κοινωνία με τις μειονότητες, με τις θρησκευτικέ μειονότητες, με όλο το ιστορικό υπόβαθρο. Και επίσης κάτι που θα πρέπει πολύ συχνά να τονίζουμε. Είναι οι συστάσεις και οι κατευθυντήριες γραμμές για τις θρησκευτικέ ελευθερίες. Στην προηγούμενη θητεία της Επιτροπής μας ασχοληθήκαμε με τις κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και είδαμε πόσο σημαντικές είναι αυτές για τις σχέσεις μας με τις τρίτες χώρες. Με οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Έχουμε μερικά μέσα και εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και καλά θα κάναμε να τα χρησιμοποιούμε, αλλά πολύ συχνά αυτά τα χρησιμοποιούμε κατόπιν εορτής. Όταν τελειώσει η ένοπλη σύραξη, κατά τη διάρκεια της σύραξης, είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσεις αυτά τα μέσα, τα πολιτικά που έχει στη διάθεσή σου. Θα πρέπει λοιπόν να ασκήσουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη επιρροή σε όλους τους γνωστούς ε, και με όλους τους διάβλους που έχει ο καθένας για να τερματιστεί η βία. Γιατί η κλιμάκωση της βίας και της σύγκρουσης και του πολέμου είναι κάτι το οποίο έχει αδιανόητες συνέπειες. Και ωραία είναι να συζητάμε διάφορα πράγματα, αλλά ακόμα καλύτερα να τα τακμηριώνουμε με στοιχεία, με γεγονότα. Γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου, όλα αυτά θα πρέπει να στοιχειοθετούνται από τη διεθνή κοινότητα. Γιατί αργότερα θα έρθει έτσι η συμφιλίωση. Αλλιώς δεν μπορεί να λογοδοτεί κανείς. Υφίσταται τόσο αδυνά, τόσε ζημίε, τόση συμφορά όλε αυτέ οι κοινότητε, χριστιανικές και άλλες. Έχει δηλώσει το Ισλαμικό κράτος ότι θέλει να τους εξαφανίσει από την περιοχή. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, αλλά το σημαντικότερο είναι η καλή βούληση. Ε, σας υπόσχομαι ότι τελειώνω. Έχουμε ε, την πρόθεση να δράσουμε και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για να βγει και κάτι από τη σημερινή ακρόαση. Όχι απλώς μια δήλωση ότι πω από τι φρικτή που είναι η κατάσταση, αλλά να δείξουμε ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε και πόσο προσιλωμένοι και δεσμεσμένοι είμαστε να δραστηριοποιηθούμε και πρόθυμοι. Ίσως να μην αρκούν τα ψηφίσματα, γιατί είναι μόνο λόγια. Ίσως θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει κάτι πιο χειροπιαστό για να δρομολογήσει αλλαγές εκεί, για να γίνει κάτι έτσι ώστε να βοηθηθούν αυτές οι διακόμενες μειονότητες, όχι μόνο εκεί, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου. Ένα τελευταίο. Αν θα πρέπει να παραμείνουν στην Μέση Ανατολή οι χριστιανοί να φύγουν. Πού να πάνε, στην Ευρώπη? Θυμίζω έναν επίσκοπο που είχε πει πριν από δύο χρόνια ότι αν δεν υπάρχουν χριστιανοί στη Μέση Ανατολή, στο Ιράκ, στη Σύρια, τη μέρα που δεν θα υπάρχουν εκεί χριστιανοί, θα έχουν χαθεί ένα εκατομμύριο ζωές. Γιατί θα χαθεί στη συνέχεια άλλο ένα εκατομμύριο ζωές, γιατί θα ε, υπάρξει ε, μία επιθυμία για εκδίκηση. Ενώ εμείς θέλουμε τη συμφιλίωση. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε όσους διώκονται, ακόμα και τους μη χριστιανούς και τους μουσουλμάνους, είναι απαραίτητο να το κάνουμε. Και αυτό είναι από τα βήματα προς τη συμφιλίωση. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις κοινότητες και όλους τους εκπροσώπους και, και τους Συγγνώμη που με ακρηγόρησα. Ευχαριστώ. Ζητώ τη συνεργασία σας. Έχουμε 11 λεπτά μόνο. Και πολλά μέλη θέλουν το λόγο. Δύο μέλη. Ο κύριος Όλβενη. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και θα είμαι σύντομος. Ε, αν ξεπεράσω τα τρία λεπτά, κάντε μου νόημα. Για μέχρι πριν από δύο εβδομάδες ήμουν στο Ιράκ και μάλιστα πέντε φορές τα τελευταία χρόνια. Ίσως καλό θα ήταν να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα για να είμαι πιο σαβή στα, ου... στα Ουγγρικά. Ευχαριστώ. Ξέρετε λοιπόν, έχω πάει στη Τσετσενία στους κόλπους μιας οργάνωσης και δεν είμαι μόνο εκπρόσωπος των, στην πολιτική σκηνή της χώρας μου. Έχω υπάρξει επιτόπου, έχω δράσει επιτόπου. Μπορώ να σας πω πάρα πολλές ιστορίες για όλα αυτά τα θέματα και ξέρω πολύ καλά τι πρέπει να γίνει. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που μίλησαν πριν από μένα η απουσία εκπαίδευσης, η απουσία σχολείων, η ανεργία, αυτά είναι τα τεράστια προβλήματα. Η Ευρώπη δεν καταλαβαίνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες ε, παιδιά δεν έχουν σχολείο να πάνε. Εάν δούμε τι έχει γίνει στη Τσετσενία, σε έξι μήνες έχτισαν οχτώ σχολεία. Άρα ο κόσμος που δουλεύει επί τόπου, οι οργανώσεις, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις μπορούν να δράσουν γρήγορα εάν τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθήσει αυτού τους ανθρώπους και δεν υψώσει ε, γραφειοκρατικά εμπόδια. Αυτό πρέπει να το πούμε. Οι τοπικές οργανώσεις δεν γνωρίζουν απαραίτητα ε, τι είναι αυτό το οποίο θα λάβουν. Έχουμε εξαιρετικούς επικεφαλείς ε, στο, στις ΜΚΙΟ και θα πρέπει να είναι σε επικοινωνία η μία με την άλλη, γιατί δεν γνωρίζει ε, η μία τι θα πράξει η άλλη πολύ συχνά. Ξέρετε, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις επίσης δεν είναι μακριά, ε, δουλεύουν εκεί επί τόπου και πρέπει να κάνουμε διάλογο με αυτούς, με εκείνες. Επιτρέψτε μου, ε, κυρία Πρόεδρε, επίσης να πω το εξής. Έχει δίκιο ο συνάδελφος Τάνοκ όμως ας δούμε λίγο το μέλλον. Έχω την εντύπωση ότι οι χριστιανοί είναι στη θέση των μειονοτήτων, αν θέλετε, ή των ευπαθών ομάδων του, ε, κατά τη διάρκεια των κομμουνιστικών καθεστώτων ή κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 ενίοτε σε ορισμένα μέρη. Δηλαδή, δεν μπορεί να ακουστεί τόσο η φωνή τους. Θα πρέπει να μετράνε αυτοί οι άνθρωποι, να μετρούν, να έχουν σημασία, να υπάρχουν, να είναι υπαρκτοί, να είναι παρόντες. Δεν μπορούμε να λέμε ότι όλοι έχουν το, την ίδια σημασία και τελικά να μην την έχουν. Θα πρέπει να πούμε ε, ξεκάθαρα ότι οι άνθρωποι αυτοί μετρούν για την Ευρώπη. Σωστό να πούμε ότι ναι, βοηθάω και τους μεν, βοηθάω και τους δε, εγώ ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να το πω έτσι. Ωστόσο, να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε και προσωπική ευθύνη εναντί των χριστιανών. Είναι και πολιτιστική, πολιτισμική μας ευθύνη εμάς εδώ στην, ε, στην Ενωμένη Ευρώπη. Και θα πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε αυτή η χριστιανική παρουσία 2.000 ετών και πλέον να παραμείνει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ας μην γινόμαστε γελοί, ας είμαστε σοβαροί. Είπα τρία λεπτά ότι θα μιλήσω, δώστε μου άλλο ένα παρακαλώ. Να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ ξέρω τι μπορώ να κάνω εδώ. Τι μπορεί να κάνει η κυρία Μογκερίνη στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ο καθένας δηλαδή να ασχοληθεί με το φάκελό του, με το θέμα του και ο καθένας να διεκδικήσει από τους ανώτερους του και από την κυβέρνησή του βοήθεια, γιατί χι χρήματα θα βοηθήσουν ψη οικογένειες. Μπορούμε να φιλοσοφούμε να φιλοσοφούμε ε, ατερμόνος και ασταμάτητα, αλλά ε, βασικά για τη χρηματοδότηση είναι η συζήτηση. Αναπτυξιακή βοήθεια. Ας συνέλθουμε γιατί αλλιώς θα ντρεπόμαστε για αυτά τα οποία δεν θα έχουμε καταφέρει να κάνουμε. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ ο κύριος Ντέμες Μέκερ, ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, θα μιλήσω Ολλανδικά και θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απολύτως με, το, ε, με τα σχόλια του Ούγκρου συναδέλφου που μίλησε πριν από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, εκπροσώπους, τους ομιλητές για τις παρεμβάσεις τους, για τις παρουσιάσεις τους. Πράγματι ήταν εξαιρετικά σημαντική η διοργάνωση αυτής της ακρόασης. Ε, ήταν μια πρόταση η οποία με ενθουσίασε εξ αρχής, αμέσως μόλις έλαβα την πρόσκληση. Μπορεί το θέμα να είναι πραγματικά ζωφερό, όμως η διοργάνωση της ακρόασης είναι εξαιρετικά σημαντική. Τα δικαιώματα των μειονοτήτων, οι ελευθερίες, το καθεστώς ΔΑΕΣ είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Αυτό ξεπερνά το μυαλό μας. Ε, βλέπουμε τις πιο σκοτεινές σελίδες ιστορίας μας και θα πρέπει να καταλάβουμε τι έκταση έχει αυτή η καταστροφή. Και επιπλέον, όλος αυτός ο τρόμος και η τρομοκρατία έχει προσλάβει και μια νέα διάσταση με την επαγγελματική προπαγάνδα που κάνουν και στο ίντερνετ, ε, στα μέσα κοινωνική δικτύωση, στο παγκόσμιο δίκτυο. Και ε, αυτή η ε, κατάπτυστη ιδεολογία βρίσκει τέτοια διάδοση που αγγίζει τους δικούς μας ανθρώπους και τους μιλάει. Η έκθεση αυτή είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή, αξίζει να διαβαστεί. Κανονικά θα πρέπει να διαβάζεται υποχρεωτικά από όλους όσοι ασχολούνται. Είναι πολύ ε, συνοπτική. Ε, και εγώ συγκρατώ κυρίως ότι υπάρχει ανάγκη ε, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι διεθνείς οργανισμοί Ευρωπαϊκή Ένωση να τεκμηριώνονται ποιες είναι οι μειονότητες που έχουν μπει στο στόχαστρο και να ε, φροντίσουμε και οι αρχές, οι κρατικές να ε, τηρούν ένα μητρό ε, αγνοωμένων για ψυχοκοινωνική υποστήριξη, γιατί πρόκειται για οικογένειες, για κοινωνίες που υφίστανται τεράστια βία. Συμφωνώ ότι θα πρέπει από τώρα διεθνώς να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα διαμορφωθεί, πώς θέλουμε εμείς να οργανώσουμε την εποχή μετά το Ισλαμικό κράτος. Τα προβλήματα θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν σε διάφορες περιοχές. Γι' αυτό ο κόσμος που έχει εκδιωθεί θα πρέπει να γυρίσει σε ασφαλή συστήση. Και δεν έχω καταλάβει τι γίνεται με τη γεωπολιτική πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή. Ε, έχει αλλάξει η κατάσταση σε σχέση με 10 χρόνια πριν. Ε, δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα υπάρχει θέση για τους Κούρδους, ας πούμε, ε, που χρειάζονται νέες δομές για να μπορούν να υποδέχονται και οι τις θρησκευτικέ και άλλες. Ε, η κοινότητα θα πρέπει να προβληματιστεί για τα λάθη της και να σκεφτούμε από τώρα ένα σενάριο στο οποίο ελπίζω να έχει ιτηθεί ε, το Ισλαμικό κράτο, να έχει εκριζωθεί και να έχει εξαφανιστεί. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν και τις υποδομές, δρόμους, σχολεία, τα κτίρια αλλά και οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ του πληθυσμού. Έχει γίνει τεράστια ζημιά ήδη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να απαντήσετε σε όλα αυτά, αλλά αυτό με ενδιαφέρει πώς μπορεί καλύτερα να συνεισφέρει η διεθνής κοινότητα από τώρα για την εποχή μετά το Ισλαμικό κράτος, ιδιαίτερα για τη συμφιλίωση μεταξύ των πολιτισμών και για μέσα έτσι ώστε να υπάρχουν πιο αντιπροσωπευτικοί θεσμοί επιτόπου, κρατικές οντότητες δηλαδή. Ευχαριστώ. Έχουμε μόνο τρία λεπτά μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Και τελικά δεν μπορώ να ξαναδώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας, αλλά θα ξαναδώσω το λόγο για ένα λεπτό και θα ολοκληρώσουμε. Μάλιστα, ευχαριστώ τους ομιλητές, ευχαριστώ και σε όσους έφεραν αυτή τη συζήτηση στην Επιτροπή εδώ. Εδώ δεν μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια σε όλους, όλους τους εκτοπισμένους και σε όλες τις μειονότητες που είναι υπό τεράστια πίεση. Αλλά αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε ως πολιτικοί, ε, θα έπρεπε το θεσμικό μας όργανο να λάβει κάποιες ε, πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις. Τα προβλήματα δεν προκύπτουν από το πουθενά, δημιουργούνται από κάποιες οργανώσεις ε, και άτομα. Ίσως, Πρόεδρε, θα έπρεπε να απευθύνουμε κάποια έκκληση στην Υπηρεσία εξωτερική δράση και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες δράσεις εναντί όσων υποστηρίζουν τον, το Ισλαμικό κράτος και άλλες ενόπλες ομάδες. Δεν πιστεύω ότι εδώ μιλάμε για μυστηριώδες ομάδες και χώρες ε, που ε, υλοποιούν αυτές τις δραστηριότητες. Έτσι λοιπόν σας παροτρύνω ένθερμα να περάσουμε σε κάτι συγκεκριμένο από αυτή τη συζήτηση και να διαβάσουμε τις συστάσεις μας ε, στις αρμόδιες αρχές. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο. Σε ένα λεπτό πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλου του προσκεκλημένου και λυπάμαι που δεν σα ξαναδίνω το λόγο. Πιστεύω ότι σήμερα τι συνέβη. Είχαμε μια μισή ώρα στη διάθεσή μα ε, και κατόπιν ε, χρησιμοποίησαμε δύο ώρε από το χρόνο και δεν μπορούσαμε να σα ακούσουμε και πάλι όλου. Έτσι λοιπόν πρέπει να συμπεράνω ότι πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Επίσης, ε, ζητώ συγγνώμη από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, γιατί δεν μπορούμε να σας δώσουμε τον λόγο. Ίσως ε, στην επόμενη συνεδρίαση να σας δώσουμε το λόγο. Ελπίζω να έχουμε χρόνο. Δεν μπορώ να κάνω περαιτέρω συμπεράσματα, δεν νομίζω ότι υπάρχουν κάποια συμπεράσματα τα οποία μπορούμε να ξαγάγουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα που μας προβληματίζουν και πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη περίοδο. Απλώς θέλω να σας κάνω μια ενημέρωση όσοι ζήτησαν περισσότερη συνεργασία μεταξύ ε, ΜΑΣΡΕΚ και Υποεπιτροπής ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σήμερα έχουμε μία συνεδρίαση στις 2 η αποστολή για τις χώρες του ΜΑΣΡΕΚ και θα συζητήσουμε τα θέματα του Ισλαμικού κράτους ε, και θα είναι με την International Crisis Group, με την ομάδα για τις διεθνείς κρίσεις. Αν θέλετε μπορείτε να συμμετάσχετε στις 2 και ευχαριστώ και τους διερμηνείς για τις προσπαθίες τους. Ας συνεχίσουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ και την πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ahora a los los miembros Παρακαλώ τα μέλη του mantendremos Παρακαλώ τα μέλη του διευρυμένου Προεδρείου, μάλλον τα μέλη της Επιτροπής μας να παραμείνουν, διότι έχουμε και συνέχεια συζήτηση